Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα συνάδελφοι. Έχουν περάσει 8 λεπτά από τις 9. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Περνάμε στο σημείο 11, σύσταση στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τη Λιβύη, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Να ρωτήσω τον κύριο Αντζέρι, όχι, δεν θέλει να πάρει τον, ε, τον λόγο. Οπότε μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Ξεκινάμε λοιπόν. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική... Ε, η τροπολογία, συγγνώμη, 86 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 105 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία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 κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καλύτερα να το ελέγξουμε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά Ψηφίζουμε λοιπόν επί της τροπολογίας 151 ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 13 ψηφί, υπέρ, 32 κατά. Απορρίπτεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 162 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 164. Έλεγχος. Ελέγχουμε την τροπολογία 162 της κυρίας Λόχ Μπίλερ, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Three colleagues missing, two colleagues missing, one colleague. Να ψηφίσουν όλοι παρακαλώ. Πέρας πληροφορία, 10 υπέρ, 22 κατά, 15 αποχές. Απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 168 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 169 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές Εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε την 170. Ωραία. Να ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 170. Άρχεται η ψηφοφορία. It's Πέρας. Εγκρίνεται. 171 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 172 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Να ελέγξουμε την τροπολογία 172. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε παρακαλώ, ψηφίστε τώρα. Πέραση ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 173 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πάμε σε τολογικές σκέψεις. 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ψηφίζουμε επιστημολογική σκέψη 8. Ψήφιστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 27 ψήφου υπέρ, 21 κατά. 9 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε. Ψηφίστε παρακαλώ για το 9. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ με την κάρτα σας. closed. Πέρας, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Καλύτερα να, να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας είμαστε καλύτερα σίγουροι. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται, μάλιστα. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε στο 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 η, τροπολογία της μέρας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 35. Γιατί 34 θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Κανένα πρόβλημα. Ψηφίστε παρακαλώ για τα 34 ηλεκτρονικά. Πέρας, 21, 27 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε. Κανένα πρόβλημα. 37. Αν και νομίζω ότι ήταν ε, σαφής η διαφορά, αλλά εν πάση περιπτώσει ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Ε, 4 υπέρ, 40 κατά. Ποιο ζήτησε έλεγχο τώρα ονομαστική ψηφοφορία. Πέντε λεπτά σιωπή παρακαλώ, για τιμωρία. 37 απορρίφθηκε λοιπόν, 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά αποχέ, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 44 έλεγχο. Εντάξει, α ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 44. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας ε, συνάδελφος δεν έχει ψηφίσει ακόμα. Ψήφισε. 45 υπέρ, 4 εποχές. Συγχαρητήρια. Και περνάμε στο σημείο 12, σύσταση προς το Συμβούλιο, την ε, Επιτροπή και την ΕΕ για τις ε, διαπραγματεύσεις για τον εξοικονομισμό της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χιλής. Θέλει ο κύριος Στάνοκ να πάρει το λόγο. Θέλω να πω απλώς ότι μπορούμε να περάσουμε στην πληροφορία. Ωραία. Οπότε μπορούμε να περάσουμε ε, στην ψηφοφορία αμέσω. Τροπολογία υπαριθμών 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. αποχέ. Ηλεκτρονική επιβεβαίωση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Υιοθετείται. Εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμόν 1 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά εποχές επαλήθευση. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγοι. Απορρίπτεται. 24 κατά 22 υπέρ. 31 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ξεκινάμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ. Κατά. εποχέ, Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41. Επαληθεύουμε. Επαληθεύουμε τη 41. It's Λίγη. Ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 24 κατά 23 υπέρ. 43 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική παρθμό 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ ε, δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές, επαλήθευση. Για το δεύτερο τμήμα, τις 56. It's Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική παριθμών 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά εποχέ, εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά Εποχέ. εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά Εποχέ. εγκρίνεται. 65 δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά Εποχέ. εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Εποχέ. εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά Εποχέ. εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά εποχέ, εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60, όχι, 69 κατά πίπτη. Περνάμε τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε την 6. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 24 υπέρ, 22 κατά. Συμβαστική παρελθόν 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές επαληθεύουμε την 11. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. εποχέ, Ξαναψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται και η 12. 13. Υπέρ. Κατά. Εποχέ. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά εποχέ απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά εποχέ απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά εποχέ απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά εποχέ εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 45 ψήφοι υπέρ και 3 αποχές. Συγχαρητήρια Charles. Περνάμε στο σημείο 13. Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή της Επιτροπής ΑΦΕΤ στη Μολδαβία και την Ουκρανία.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 So, half past nine. 9.30 λοιπόν συνάδελφοι. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησία διάταξή μα. Ενημέρωση σχετικά ε, με την αποστολή της Επιτροπής ΑΦΕΤ στη Μολδαβία και στην Ουκρανία 2 με 6 Απριλίου. επικεφαλής στην αντίστοιχη για η Ιαπωνία και Νότια Κορέα. Η κυρία Μισλακινέν ήταν στη συγκεκριμένη με έξι μέλη της ΑΦΕΤ και επιπλέον προσθέθηκαν στην αντιπροσωπεία μας και συνάδελφοι από την Επιτροπή του Προπολογισμού και από άλλες επιτροπές. Ευχαριστώ. Παρακαλώ την επικεφαλής να μιλήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή την αφορά στην αποστολή της Επιτροπής ΑΦΕΤ στη Μολδαβία και στην Ουκρανία. Στόχος ήταν να τροφοδοτήσουμε την Επιτροπή μας σε σχέση με τη Συμφωνία Σύνδεσης και τα αντίστοιχα έγγραφα και τις άφορες άλλες συμφωνίες που έχουμε με Μολδαβία και Ουκρανία. Όπως επίσης και η παροχή μακροοικονομικής βοήθειας σε αυτές τις περιοχές. Επίσης θέλαμε να αποτιμήσουμε την περίπλοκη πολιτική κατάσταση εν ώψη σημαντικών επερχόμενων εκλογών. Όπως είπατε και εσείς Πρόεδρε, είχαμε με έξι μέλη της ΑΦΕΤ στην αποστολή αυτή, ο κύριος Γκάλερ ο εισηγητής, ο Στραβίτσιους, Φραντσούλικα, Χέλμουτ Σόλτς, και ο κύριος Ντάριους Δρασάιτε από την αντιστοιχή Επιτροπή για τη Μολδαβία. Είχαμε επίση και συναδέλφου από την Επιτροπή Προπολογισμού και από τι Διακοινοβουλευτικέ Επιτροπέ. Είχαμε ένα πολύ έντονο και γεμάτο πρόγραμμα. Είχαμε πολλέ συναντήσει, δύο συνδεύξει τύπου και επισκέψει επιτόπου. Και στη Μολδαβία και στην Ουκρανία συναντήσαμε τους πρωθυπουργούς, τους κυβερνητικούς εκπροσώπους, τους ε, πρόεδρους, τους προέδρους των Επιτροπών Εξωτερικών Παθέσεων των Κοινοβουλίων, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, πρεσβευτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Επιπλέον, στην Μολδαβία συναντήσαμε και τον Πρόεδρο και πήγαμε να επισκεφτούμε προγράμματα που, χρηματοδο... που χρηματοδοτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιστέρια συγκεκριμένα. Εκεί τονίστηκαν θέματα τα οποία αφορούν είναι ειδικινού ενδιαφέροντος και διάρκεια τη ε, αποστολή μα και ιδιαίτερα να αναφερθώ για τη Μολδαβία. Εμεί υποστηρίξαμε την εφαρμογή τη συμφωνία ε, Σύνδεση και τονίσαμε την ανάγκη ε, πρόοδο όσον αφορά τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου και την πρόσφαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πάρα πολλέ συζητήσει επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση τη διαφθορά και στην ανάγκη αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη διερεύνηση τραπεζικών απατών. Κύριο στοιχείο εδώ είναι οι μεταρρυθμίσεις. Ο κύριο Στραβίτσιος βεβαίω θα σα ενημερώσει λεπτομέρεστερα για αυτά τα θέματα. Εκλογέ συζητήθηκαν επίση λόγω των επερχομένων τοπικών εκλογών το Μάη και τι κοινοβουλευτικέ στο τέλο του έτου. Πρέπει να σα αναφέρω ότι λάβαμε διάφορα, δεχτήκαμε διάφορα παράπονα όσον αφορά την εκλογική νομοθεσία, πρόσβαση στα ΜΜΕ και στην πανενόχλωση κάποιων εκπροσωπών της αντιπολίτευση. Κάποιοι ανησυχούν για την εξαγωγή αυτών των εκλογών και ήδη υπάρχει σύσταση να αποσταλεί από το Κοινοβούλιο ένα, μια ομάδα παρατηρητών όπως είχε γίνει στην Ουκρανία το 2014. Τέλος, για τη Μονταβία, επικοινωθήκαμε στην εργασία του Κοινοβουλίου και ζητήσαμε από τους συναδέλφους μας να ευθετήσουν σύντομα το νέο κώδικα για τα ΜΜΕ που έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης στηρίξαμε τις προσπάθειες για ανάπτυξη νέου κώδικα διοντολογίας και κανονισμών που θα βελτιώσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο Κοινοβούλιο, στην Ουκρανία τώρα. Και πάλι στηρίξαμε την ε, εφαρμογή της συμφωνία Σύνδεσης και τονίσαμε την ανάγκη για σημείωση πρόοδος όσον αφορά τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Επίσης, επενέσαμε τις ε, τρέχουσες ε, μεταρρυθμίσεις παρά τις ε, ρωσικές επιθέσεις και επίσης τονίσαμε ότι αυτή η σύραξη θα πρέπει να ξεχαστεί. Όπως κάναμε και στη Μολδαβία, επικεντρώσαμε τις συζητήσεις στην ανάγκη για την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και επ' αυτού σχετικά η θέσπιση υψηλ... ανωτά του δικαστηρίου καταπολέμησης διαφθοράς αποτελεί μια προτεραιότητα. Φέτος τον Μάιο ή τον Ιούνιο θα γίνουν εκλογέ παρά την αντίθεση που υπάρχει από πολλού βουλευτέ στο Κοινοβούλιο και σε σχέση με τι ε, υποχρεώσει των ε, ακτιβιστών για υποβολή δηλώσεων. Ε, το συζητήσαμε και αναφερθήκαμε σε αυτό. Επίσης συζητήσαμε την μακροοικονομική οικονομική αρρωγή που παρέχει η Ένωση στην Ουκρανία και θα αφήσω το θέμα αυτό στον κύριο Γκάλου να το συζητήσει, να το παρουσιάσει εκτενέστερα. Επίσης μιλήσαμε για τον εκλογικό νόμο. Όπως έχουν πει και άλλα όργανα όπως η Επιτροπή της Βενετίας και έχουν υποβάλει συστάσεις, η διεξαγωγή όλων των μορφών εκλογών θα πρέπει να εναρμονιστεί. Αυτό πρέπει να αφορά όλες τις εκλογές. το σχέδιο εκλογικού νόμου είχε επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο τον περασμένο Σεπτέμβριο και θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό. Σε γενικέ γραμμέ θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντα ότι θα πρέπει να ευχαριστήσω του πρεσβευτές της Ένωση και τις ομάδες τους που παρήχαν θαυμάσια στήριξη σε αυτή την αποστολή πριν, κατά διάρκεια και μετά τη διάρκεια τη, όπω επίση μα παρήχαν πολύ χρήσιμε συμβουλέ επιτόπου. Και κυρίω ε, βεβαίω θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό μα τη ΑΦΕΤ για την θαυμασία δουλειά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you, Ευχαριστώ, κύριε Ανδρικίνε. Θέλουν άλλοι συμμετέχοντε στην αποστολή αυτή να τοποθετηθούν. Ο κύριος Μιχαήλ Γκάλερ έχει το λόγο. Πρώτα πήγαμε στην Μολδαβία βέβαια, αλλά όπως, όπως θέλετε πρόεδρε. Ποιος θέλει να ε, τοποθετηθεί, να πει κάτι για την ε, Μολδο, Μολδαβία. Ευχαριστώ που μου, δίνετε και πάλι το δικαίωμα λόγου. Ο κύριος Αστρεβίτσης. Πραγματικά ήταν εξαιρετική η επίσκεψη αυτή στην Μολδαβία. Ήταν ε, πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά μας. Ε, είχαμε μαζί μας ε, και τον κύριο Μουρεσάν από την Επιτροπή Προπολογισμών. Είχαμε πραγματικά πάρα πολλές ε, συναντήσεις με κρατικούς αξιωματούχους, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με μονομενούς πολιτικούς. Και για να είμαι ειλικρινής, υπάρχει μια κάποια διαφωνία σε διάφορα θέματα ανάμεσα σε εμά και του κρατικού αξιωματούχου της Μολδαβία και δεν υπάρχει λόγο να το κρύψουμε. Και εγώ θα χώριζα τα θέματα ε, σε δύο κατηγορίε: Οικονομικά θέματα, εμπορικά θέματα, ε, αφενός και αφετέρου πολιτικά, δικαστικά ζητήματα, ζητήματα που συνδέονται με το κράτο δικαίου. Στην ε, οικονομική πλευρά τα πράγματα είναι θετικά οι εμπορικές συναλλαγές αυξάνονται, ε, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικεντρωθούμε στις οικονομικές εξελίξεις στη Μολδαβία, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την ε, βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος. Από πολιτικής πλευράς όμως και δικαστικής υπάρχει μια έντονη αίσθηση διαμάχης ε, ή εν πολλά ανοιχτά θέματα ε, καθώς ε, θα εφαρμοστεί και ο εκλογικός κώδικας που αποφασίστηκε το φθινόπωρο στις εκλογικές διαδικασίες στην Μολδαβία και θεωρούμε ότι δεν πρόκειται για θετική εξέλιξη στη χώρα αυτή και ελπίζουμε να υπάρξουν ευκαιρίες έως τότε οι Μολδαβοί πολιτικοί να τροποποιήσουν τις διατάξεις αυτού του εκλογικού κώδικα πριν από την διεξαγωγή των εκλογών. Έγινε μια ανοιχτή συζήτηση για αυτό το θέμα με ε, υψηλότητα τους ε, αξιωματούχους και δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε συμφωνία από την πλευρά τους όσον αφορά την τροποποίηση αυτού του εκλογικού κώδικα. Στην δικαιοσύνη προσβλέπουμε στην πρόσληψη δικαστών και επαρκούς προσωπικού ε, στα δικαστήρια αυτά στη Μολδαβία ε, με νομικούς, δικηγόρους δικαστές και θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία αυτά τα νέα δικαστήρια το συντομότερο δυνατό και υπάρχουν κάποιες ε, περιστάσεις που επίσης μας ανησυχούν γύρω από αυτό. Τέλος, για τη διερεύνηση της τραπεζικής απάτης που είναι ύψη τη σημασίας ζήτημα και για την ίδια τη Μολδαβία και για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για τους πιστωτές, για τους δανειστές. Ε, υπάρχουν πληροφορίες που πρέπει να αποκαλύπτονται και όποτε εντοπίζονται παρατυπίες ή παρανομίες να διώκονται. Υπάρχει επίσης ένα ακόμη ζήτημα γεωπολιτικού χαρακτήρα. Υπάρχουν γεωπολιτικές, γεωπολιτικού χαρακτήρα συζητήσεις ε, ακόμη και σε επίπεδο ε, υψηλόβαθμων ε, αξιωματούχων στη χώρα, το οποίο δεν μπορώ να, τις οποίες δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ με όρους ορθού λόγου. Εντάξει, το, τα θέματα αυτά ε, εναπόκεινται βεβαίως στους αρμόδιους πολιτικούς της Μολδαβίας, αλλά παρόλα αυτά και εμείς πρέπει να παρακολουθούμε στενά τη συζήτηση αυτή. Γενικά, η επίσκεψη αυτή μας προσέφερε πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον υλικό για την ε, κοινή έκθεση που θα συντάξουμε για τη Μολδαβία και θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς κύριε Πρόεδρε που ζητήσατε από την ΕΕΔ τις επικαιροποιημένες σχετικές πληροφορίες. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν γιατί νομίζω ότι αυτές οι πληροφορίες θα διευκολύνουν και το εν γέννη έργο μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι για την ε, Μολδαβία. Κρίστιαν Πρέντα, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχες στην επίσκεψη αυτή, στην αντιπροσωπεία. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να πω δύο λόγια. Πριν την αναχώρηση της αντιπροσωπείας αυτής, μου είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι οι άλλες πολιτικές ομάδες εκτός του ΕΛΚ θα συμφωνούσαν να ψηφίσουμε ψήφισμα το οποίο είχαμε προετοιμάσει ήδη το Σεπτέμβρη. Επί τη βάση των, της δουλειάς που θα έκανε η αντιπροσωπεία στη Μολδαβία. Με έκπληξη όμως είδα την περασμένη εβδομάδα και να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποίησε και ο εισηγητής, είδα λέω με έκπληξή μου ότι αποφασίσαμε να κλείσουμε τα μάτια μας. Με την εξαίρεση του ΕΛΚ, όλες οι άλλες πολιτικές ομάδες απέρριψαν την ιδέα να εκδώσουμε ψήφισμα που θα κάνει λόγο για την κατάσταση στη Μολδαβία. Λαμβάνοντας υπόψη και τα πορίσματα της επίσκεψής μας. Η απόφαση επί για ένα ψήφισμα στο θέμα της Μολδαβίας είχε ήδη, σας υπενθυμίζω, ληφθεί το προηγούμενο Σεπτέμβρη. Πολύ κακός λοιπόν πολιτικός προγραμματισμός. Αναβάλαμε για μία ακόμα φορά την υιοθέτηση του ψηφίσματος. Η... ιδέα είναι ότι θα πρέπει να στηρίξουμε ε, μία, φιλοευρωπαϊκή συμμαχία στο Κισινιό ε, η οποία όμως δεν υπάρχει εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχει ένα κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα, που είναι μέλος της διεθνούς, Σοσιαλιστικής Διεθνούς και που έχει ακόμα την πλειοψηφία, διότι αγόρασε, πραγματικά αγόρασε τους κομμουνιστές βουλευτές του Κοινοβουλίου. Οι ολιγάρχες που ελέγχουν την ε, πολιτική ζωή στην Μολδαβία και δυστυχώς επηρεάζουν τα μυαλά και πολλών εδώ πέρα αγόρασαν, εξαγόρασαν τις ψήφους των κομμουνιστών βουλευτών και σκοπίμως κλείσαμε τα μάτια κύριε Σιγητά. Και ήθελα να σας το πω αυτό για να το υπογραμμίσουμε. Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής θα είναι καταστροφικό. Και στις επόμενες εκλογές θα κερδίσουν οι σοσιαλιστές, ο Ντοντών. Οι σοσιαλιστές είναι ακόμα χειρότεροι για από τους κομμουνιστές. Οι σοσιαλιστές είναι με τη Μόσχα. Ε, οι κομμουνιστές τουλάχιστον ήταν με τους ολιγάρχες. Ευχαριστώ πολύ που κλείσατε τα μάτια λοιπόν. Ευχαριστούμε Κριστιαν. Θα ήθελε κανείς άλλο το λόγο για τη Μολδαβία. Ωραία. Ταξιδεύουμε λοιπόν από τη Μολδαβία στην Ουκρανία κύριος Γκάλερ για την επίσκεψη εκεί. Όπως ε, θα ήθελα καταρχήν πριν πάμε στην Ουκρανία να στηρίξω όσα είπε ο κ. Πρέντα. Εκεί έχουμε έναν που φέρεται στα ελληνιστικά και κατά τα άλλα κρατάει τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα χέρια του. Και δεν φορά μόνο το κοινοβούλιο της Μολδαβίας και οι δήμαρχοι. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές κέρδισαν πάνω από 200 δήμους και ξαφνικά έχουν βρεθεί στους 600 χωρίς να έχουν ξαναγίνει εκλογές. Αυτό είναι το Δημοκρατικό Κόμμα. Εκφοβίζουν ενδεχόμενους ε, ε, υποψήφιους άλλων κομμάτων κλπ. Το γνωρίζουμε. Και στείλαμε το μήνυμα αυτό στον πρόεδρο του κόμματος. Δεν είναι σωστή αυτή η συμπεριφορά του εκφοβισμού στο δημόσιο τους ε, απειλούν ότι θα υπάρξουν, θα γίνουν αντίπεινα, στο ιδιωτικό τομέα τους απειλούν ότι έχετε φοροδιαφύγει οπότε θα σας διώξουμε γι' αυτό. Και εδώ είναι κάποιοι αυτοί που λένε ότι αγωνίζονται δίθεν εναντίον του Ντοντών και, ε, και των φίλων της Μόσχας. Δεν βλέπω μεγάλη διαφορά. Τώρα στην Ουκρανία. Και εδώ έχουμε δύσκολες αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουν οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις και πολλές, ε, πολλά κόμματα της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι πραγματικά θέλουν να γίνουν μεταρρυθμίσεις και κάποιοι άλλοι που θέλουν είτε να τις αναβάλουν τις μεταρρυθμίσεις είτε να τις ε, νοθεύσουν. Ε, η πρώτη ανάγνωση του προσχεδίου νεοκλογικού νόμου μα δίνει καταρχήν την εντύπωση ότι δεν θα περάσει από τη Βουλή, οπότε θα χαθεί ακόμα μια ευκαιρία η χώρα να αποκτήσει ένα καλύτερο εκλογικό σύστημα. Κρίμα. Υπάρχει ακόμα χρόνος βέβαια. Και αν συνοδευτεί από πολιτική βούληση μπορεί και να ψηφιστεί. Πώς είπε και η κυρία Αντρικέν ναι, κατά κάποιο τρόπο ε, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία τα έχουμε στο μυαλό μας εδώ και καιρό βρίσκονται στην ατζέντα. Δεν έχουν όμως υλοποιηθεί και γι' αυτό το λόγο η χώρα δεν έλαβε την τελευταία δόση του τρίτου προγράμματος μακροοικονομικής ενίσχυσης. 17 από τα 21 προαπαιτούμενα υλοποιήθηκαν, δεν και λίγο βέβαια, αλλά 4, 4 προαπαιτούμενα δεν υλοποιήθηκαν. Οπότε αυτά μεταφέρθηκαν στο τέταρτο μακροοικονομικό πρόγραμμα που ε, συνοδεύει την υλοποίηση της συμφωνίας με την Ουκρανία. Ε, υπάρχει και ο νόμος για το ανώτατο δικαστήριο κατά της διαφθοράς. Τροποποιεί, τροπολογίες ζητήθηκαν από την αντιπολίτευση για το πεδίο εφαρμογής και για, την, για το ποιοι θα έχουν δικαίωμα να επιλεγούν για δικαστές. Καθώς επίσης και το πώς οι δυτικοί εμπειρογνώμονες θα επηρεάζουν την επιλογή των δικαστών για αυτό το ανώτατο δικαστήριο κατά τη διαφθοράς. Δεν ψηφίστηκαν αυτές οι τροπολογίες και μας υπόθηκε ότι το Μάιο ή το, το αργότερο τον Ιούνιο θα γίνει η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου. Θα μπορούσαν να γίνει και πιο γρήγορα και θα μπορούσαν να είχαν διορθωθεί ήδη οι αδυναμίες του κειμένου. Και εδώ όμως έχουμε ε, συμφέροντα τα οποία ε, προφανώς δεν θέλουν να δουν ένα ε, αποτελεσματικό δικαστήριο κατά της διαφθοράς. Σε ό,τι αφορά τις ε, ηλεκτρονικές ε, φορολογικές δηλώσεις, πολύ καλό βήμα, διότι αυτό αποκάλυψε, ανάγκασε πολλούς ε, αξιωματούχους, κρατικούς αξιωματούχους να δηλώσουν τα εισοδήματά τους και τα χρέη τους. με πνεύμα εκδίκησης, έτσι το βλέπω εγώ, Ε, ζήτησαν να εφαρμοστεί αυτό και για τα μέλη των μη κυβερνητικών οργανώσεων που μάχονται κατά της διαφθοράς. Ε, εδώ δεν το θέμα αυτό δεν έχει σχέση με το κατά πόσον οι μη κυβερνητικέ οργανώσει θα πρέπει να είναι διαφανείς και να αποκαλύπτουν από το, τα, τις πηγές των εσόδων τους. Δεν μιλάμε γι' αυτό, μιλάμε για τα πρόσωπα τα οποία εργάζονται για αυτές τις μη κυβερνητικές και προσπαθούν να αλλάξουν την κατάσταση και να διορθώσουν το πρόβλημα της διαφθοράς. Η... Ε, το θέμα αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί. Μας βεβαίωσαν ότι θα αντιμετωπιστεί, έτσι μας είπε πάνω από το γραφείο του Πρόεδρου και από αλλού. Ε, είναι προφανώς όμως ότι το θέμα αυτό ε, βλάπτει τα συμφέροντα κάποιων συγκεκριμένων ατόμων. Οπότε αυτό είναι κάτι θετικό, ας μην εστιάζουμε μόνο στις αδυναμίες. Σε τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα, σίγουρα οι αρχές ε, έχουν πολύ περισσότερα χρήματα. και μερικές περιπτώσεις δεν ξέρουν καν πώς θα τα δαπανίσουν σωστά γιατί τώρα πια υπάρχουν περισσότερα νομικά μέτρα ελέγχου των δαπανών, οπότε κάποιοι τοπικοί αρχόντες φοβούνται μήπως κάνουν κανένα λάθος και δεν δαπανούν καν τον προϋπολογισμό τους και ε, τα νέα ποσά τα οποία προέκυψαν από την ε, αποκέντρωση. Και είναι σημαντικό να ε, επενεθούν και αυτοί οι οποίοι πραγματικά δουλεύουν καλά και δαπανούν τα χρήματα προς όφελος του πληθυσμού τους. Η μεταρρύθμιση της υγείας με πολλές ιδιωτικοποιήσεις και άλλα μέτρα πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Οπότε είμαι σίγουρος ότι η χώρα είμαι πεπισμένος ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και μην ξεχνάμε ότι ακόμα πολεμούν στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Και δαπανούν ε, μεγάλο ποσό του ΑΕΠ τους εκεί. Θα μπορούσαν όλα αυτά τα ποσά να χρησιμοποιηθούν προφανώς για... Ε, άλλες ανάγκες της οικονομίας. Ε, δεν είναι μια παγωμένη σύγκρουση. Κάθε μέρα χάνουν τη ζωή τους άνθρωποι. Ε, γίνεται πολεμάνε οι άνθρωποι εναντίον των Ρώσων ή των, αντι... αντιπροσώπων των Ρώσων. Ε, ο αγώνας γενικά στη χώρα είναι δύσκολος ελπίζουμε ότι θα βρεθούν οι κατάλληλες πλειοψηφίες έτσι ώστε να διορθωθούν όλες οι αδυναμίες που έχουν ε, εντοπιστεί και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Επιτροπή της Βενετίας κλπ. Αυτή τη στιγμή ε, νομίζω ότι υπάρχει ε, ένας εκπρόσωπος εδώ σήμερα κιόλα και θα δούμε που βρισκόμαστε. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστώ. Κύριε Γκάλερ, μήπως κάποιος άλλο θα ηθελε να προσθέσει τίποτα μετά από αυτά που ακούσατε για την Ουκρανία. Ποιο του κύριε. Συνάδελφοι, Πρόεδρε, θα ήθελα να πω τα εξής. συχνά μιλάμε για τον Όρμπαν και τον εθνικισμό. Αλλά για την Ουκρανία εγώ είμαι της άποψης ότι η ζυγαριά αρχίζει να γέρνει υπέρ των εθνικιστών στην Ουκρανία. Δεν ξέρω κατά πόσο τα μέλη της αντιπροσωπείας ε, μίλησαν για την νομοθεσία η οποία αφορά τις διακρίσεις κατά μειονοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα και στη χρήση της γλώσσας. Εγώ ως Ούγγρος μπορώ να σας πω ότι όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ουγγαρία αυτό απειλείται και αυτό νομίζω ότι δεν επιτρέπει στις ε, μειονότητες των Ούγγρων να επιβιώσουν. Οπότε γίνεται ακριβώς με αυτό το θέμα το, ε, της εκπαίδευσης όσον αφορά τους Ούγγρους. Okay, thank you, Ευχαριστώ. Ο κ. Γκάλερ θα ήθελε να απαντήσει αμέσω. Ναι, βεβαίω Το αντιμετωπίσαμε αυτό το θέμα και το συζητήσαμε. Και είπαμε ότι στους εφαρμοστικούς νόμους θα σεβαστούν πλήρως τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας της περσμένης εβδομάδα και της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και είπαμε στη διατύπωση ακριβώς fully implement πλήρης εφαρμογή σε σχέση δηλαδή με το χρονοδιάγραμμα το οποίο είχε αναβληθεί. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια δικαιολογία αυτή τη στιγμή για το αντίθετο. Ώστε δηλαδή αυτό που θα εφαρμόσουν να είναι αντίθετο με αυτά που λέει η Επιτροπή της Βενετίας ή αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την εκπαίδευση των μειονοτήτων. Αυτό νομίζω πρέπει να το αναγνωρίζουν όλοι. Θα πρέπει να συνεχίζεται πάντω, να συνεχιστεί πάντων ο διάλογος με όλε τι ενδιαφερόμενες χώρες μέλη. Διάλογος ο οποίο, όπως είπα, συνεχίζεται και νομίζω ότι η κατάσταση θα εξελιχθεί ομαλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. άλλε παρατηρήσεις. Όχι από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ τον Άιμαρ και την ε, και τους υπόλοιπους για αυτή την ενημέρωση. Θα μπορούσαμε τώρα να πάμε κατευθείαν στο 14, σημείο της ημερησίας, ενημέρωση σχετικά με την αποστολή στην Ιαπωνία και στην Νότιο Κορέα, 2 με 6 Απρίλη. Αυτή η αποστολή στις δύο έγινε από τις 3 μέχρι τις 6 του Απρίλη. Είχατε τιμή να αυτής της αποστολής Είχαμε 8 μέλη, Ράφκα και Μπρόκα από το ΕΛΚ, Σφίτσα, από, το, από τους Σοσιαλιστές, Πάσχο επίση, από το ECR ε Σανέσκι από την Άλντε, Ορμα και από τους Πράσινους ο Κλάνς Μπουχνέρ. Κίνητρο μας ήταν να δείξουμε, να δώσουμε στήριξη στους σταδικούς μας εταίρους στην Κορέα και στην Ιαπωνία, γιατί είναι οι πιο στενοί μας εταίροι στην περιοχή αυτή και έχουν τις πιο μακροχρόνιες σταθερές δημοκρατίες στην περιοχή αυτή. Είχαμε και τη στρατηγική συμφωνία με την Ιαπωνία και την οικονομική συμφωνία, η οποία θα πρέπει να, οι οποίες θα πρέπει να υπογραφούν στην επόμενη διάσκεψη κορυφής ΕΕ Ιαπωνίας, που ελπίζω θα γίνει εδώ στις Βρυξέλλες του Ιούλιο. Και μετά ελπίζουμε βέβαια το Συμβούλιο θα παραπέμψει τις ε, συμφωνίες αυτές τρεις μέρες αργότερα και μετά θα συγκληθεί η ΑΦΕΤ ώστε να τις εγκρίνει και θα ψηφιστούν κατά τη διάρκεια της θητείας μας στην Ολομέλεια εισηγητής και ο Πίτελε. Επίσης, εξίσου σημαντικό ήταν το να εξετάσουμε ακριβώς τις βαλιστικέ πυρηνικέ δοκιμέ που κάνει η Βόρεια Κορέα και να δούμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να συμβάλλει σε μια διαρκή ειρήνη και στην αποπυρηνικοποίηση τη Χερσονήσου. Θέλαμε επίση να στηρίξουμε τις ε, νέες, τις πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά το ενδεχόμενο υψηλού επίπεδου επαφών με τη Βόρεια Κορέα και για το ρόλο μα όσον αφορά τι ειρηνευτικές διαδικασίε και συνομιλίες ε, θέλαμε να είμαστε όχι ένας μεσολαβητή, αλλά ένα διευκολυντής ώστε να αντιμετωπιστεί σωστά αυτή η κρίση. Κάποιες χώρες μας έχουν πρεσβείε στην Πιόν Γιάνγκ και συνεχίζουμε τις επαφές με όλου τους ε, ενδιαφερόμενου, συγκεκριμένα βέβαια είπα και την Βόρειο Κορέα. θα μπορούσαμε βεβαίως να προσφέρουμε την φιλοξενία αυτών των συνομιλιών υψηλού επίπεδου, αλλά ταυτόχρονα βέβαια θα πρέπει να συνεχίσουμε μια ανυποχώρητη πολιτική μέχρι να δούμε αυτά αποτελέσματα στην αποπυρηνικοποίηση, την, ε, την απάλληψη των πυρηνικών όπλων και τον αφοπλισμό. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι έτοιμη να στηρίξει την εφαρμογή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας. Αυτά από τη δική μου πλευρά. Είχε διοργανθεί πολύ καλά η αποστολή μας και να ευχαριστήσω τις αντιπροσωπείες μας σε Σεούλ και Τόκιο και τη γραμματεία μας επίσης. Αυτά από μένα δεν ξέρω αν έχετε να πείτε εσείς τον Μπράφκα. Ευχαριστώ, Ντεβίτ. Να μην τα επαναλάβω και εγώ. Είχε διοργανωθεί πολύ καλά αυτή η αποστολή. Το σημαντικότερο κατά την άποψή μα ήταν ότι αυτή η αποστολή ήταν πραγματικά κέρια. Θα έχουμε και διάσκεψη κορυφή όπω είπαμε τον Ιούλιο εδώ στι Βρυξέλλε. Αλλά είχαμε και το θέμα τη Βορεια Κορέα. Είχαμε εξελίξει από αυτού. Όπω ξέρουμε, πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί με τις κυρώσεις, γιατί δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει μετά από τις διασκέψεις και την συνάντηση Τραμπ και Κιμ. Θα δούμε τι θα γίνει λοιπόν. Ας είμαστε αισιόδοξοι και ως Ένωση εμείς θα πρέπει να συμβάλλουμε σε μια διαρκή ειρήνη. Αυτό είχα να πω. Ήταν καλό ταξίδι πάντως και είχαμε επαφές με διάφορους αξιωματούχους, υπουργούς εξωτερικών, πρόεδρους κοινοβουλίων. Ήταν λοιπόν πολύ καλή αυτή η αποστολή και αναμένουμε με ανυπομονησία τις εξελίξεις σε αυτή την περιοχή γενικότερα, αλλά ειδικότερα στην Χερσόνησο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρος. Ευχαριστώ, κυρία Ντουμπραφιά, για τη σχόλιά σας. Επόμενος ε, ομιλητής, Ούρμας Πάετ. Ευχαριστώ. Θέλω να προσθέσω τρία πράγματα. Πρώτον, η Ευρώπη και ολόκληρο ο κόσμος πρέπει να διατηρήσει τις κυρώσεις και την πίεση που ασκείται γιατί είναι σημαντικό να δούμε αλλαγές στο καθεστώς της Βόρειας ε, Κορέας και με τα πυρηνικά αλλά και με τις ε, αποτρόπες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεχίζονται. Άρα μετά τις συνόδους ε, κορυφής που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα μεταξύ Βορρά και Νότου και τον Μάιο μεταξύ Βόρειας Κορέας και ΙΠΑ υπάρχει ένα παράθυρο ελπίδας αλλά εξακολουθούμε να μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα γιατί όταν μιλάμε για κυρώσεις οι πιέσεις αυτές συνεχίζονται να ασκούνται ε, ιδίως ε, όταν συνυπολογίσει κανείς και την παρουσία της Κίνας που, έχει, που είναι και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Κορέας. Δεύτερον, υπάρχει και μια μεταστροφή και στη Νότια Κορέα όσον αφορά την επανένωση για ε, πολλά χρόνια θεωρούσαμε ότι οι Νοτιοκορεάτες θέλουν την επανένωση. Φαίνεται όμως ότι μετά από 40 χρόνια, μετά από, ε, μάλλον οι, άνθρωποι που είναι κάτω των 40 ετών δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα επηρεάσει το μέλλον της Χερσονήσου. Και όσον αφορά τα, τις διμερείς μας σχέσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα, Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με, ε, στον τομέα της κυβερνοασφάλειας οι χώρες αυτές είναι και οι δύο πολύ προηγμένες στον τομέα αυτό. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες τους και να προχωρήσουμε σε μια πραγματικά πρακτική συνεργασία στον τομέα αυτό και με τις δύο χώρες, και με την Ιαπωνία και με την Νότια Κορέα. Ευχαριστώ. Ούρμα Σπάετ, θέλει κάποιος άλλος το λόγο και να πει κάτι για την αποστολή αυτή πέραν των όσων ήδη ακούστηκαν. Όχι από ό,τι φαίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Το επόμενο σημείο, το υπαριθμό 15, είναι ανταλλαγή απόψεων με τον Πρωθυπουργό της Τινησίας, ο οποίος όμως δεν έχει καταφθάσει προφανώς, οπότε λέω να αναστείλουμε τη συναδρίασή μας έως τις 10 ε, και 25 για να μπορέσουμε έγκαιρα στην ώρα μας στις 10.30 ε, να ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα. Οπότε θα κάνουμε ένα διαλυματάκι 20 λεπτών για καφέ. Bulgarien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 Κυριε and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα να συνεχίσουμε τώρα τη συνεδρία τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και να περάσουμε στο σημείο 15 τη ημέρα διάταξη. Είναι χαρά και τιμή για όλου μα να υποδεχόμαστε εδώ στην Επιτροπή μα τον αρχηγό τη κυβέρνηση τη Τινησία, τον κύριο Γιούσεφ Τσαχέντ. Καλώ ήρθατε. Μου υπόθηκε ότι... Μέρχαμπα, μέρχαμπα, έτσι λέτε στη γλώσσα σας. Σχεδόν ε, τα κατάφερα να το προφέρω σωστά. Σας ε, καλωσορίζουμε λοιπόν και να τονίσω εξ αρχής ότι τα μέλη της Επιτροπής μας παρακολουθούν στενά την κατάσταση στη Δυνησία εδώ και πολλά χρόνια για μας η χώρα σας αποτελεί φάρο της δημοκρατίας στη Βόρεια Αφρική και έχει διέλθει μια μακρά και σύνθετη διαδικασία για να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Τινησία και το γεγονό ότι η διαδικασία μεταρρυθμίσεων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Είμαι βέβαιο ότι τα μέλη τη Επιτροπή μα θα ήθελαν να μα πείτε περισσότερα στοιχεία σχετικά με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και ε, του στόχου μεταρρυθμίσεων τη κυβέρνησή σα. Θέλω επίση να τονίσω ότι μια ανοιχτή, σταθερή και δημοκρατική Ισία είναι κοινό μας συμφέρον, ωστόσο ο λαός της Τινησίας δεν αξίζει μόνο δημοκρατία και σταθερότητα, αλλά πρέπει να επωφεληθεί και από θετικέ δημόσιες πολιτικέ και καλή διακυβέρνηση. Η οικονομική ανάπτυξη ενισχύει τη δημοκρατική σταθερότητα και θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα στοιχεία για το τι κάνετε σε αυτή τη διάσταση. Επίσης, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι οι τοπικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν τελικά σε 6 Μαΐου 2018 έπειτα από μια καθυστέρηση δύο ετών και έμπρακτα ως υποστήριξη από πλευράς μας προς τη δημοκρατική διαδικασία στην Τινησία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να στείλει εκλογικούς παρατηρητές, κάτι που δεν ήθιστε σε τοπικές εκλογές. Ο κύριος Καστάλτο θα είναι επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας. Τέλος, στο πλαίσιο της μεταβατικής διαδικασίας για τη δικαιοσύνη θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα στοιχεία σχετικά με την πρόσφατη αποφάση του Κοινοβουλίου της ε, Τινησίας να μην ε, παρατείνει την εντολή της Επιτροπής ε, Αλήθειας και Αξιοπρέπειας. Χωρίς περαιτέρω χρονοτεβή, να σας καλωσορίσω, να σας δώσω το λόγο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε σε ποια γλώσσα θέλετε να μάθετε. Ε, από τις 24 που έχουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι θα μιλήσω γαλλικά. Καταρχήν, τις ευχαριστίες μου στον κύριο Ντέβιτ Μακάλιστερ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, που διοργάνωσε την συνάντηση, την κοινή τη αυτή συνάντηση. Να Πρέπει να μιλήσουμε για τον, τη διαδικασία εκδημοκρατισμού στην Τινησία, διαδικασία που ξεκίνησε το 2011 μετά την επανάσταση της 24ης Ιανουαρίου. Και να δούμε επίσης και την πρόοδο την οποία, η οποία έχει επιτευχθεί στην ε, στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Τινησίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά ε, τον εκδημοκρατισμό της χώρας ε, ε, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα. Σήμερα η δημοκρατία είναι εδρεωμένη στην την Ισία, ήταν μια μεγάλη πρόκληση αυτό για τους πολίτες μας. Έχουμε σημειώσει σημαντικές προόδους σε ό,τι αφορά την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία συνείδησης, νομοθετήματα τα οποία καθορίζουν πως η χώρα είναι ελεύθερη και δημοκρατική μέσω για... και βέβαια κυρίως το Σύνταγμα του 2014 που είναι ένα πρωτοποριακό φιλελεύθερο σύνταγμα που ε, καθορίζει και εδραιώνει τα, ε, τις ε, διάφορες ελευθερίες, έκφραση, συνείδηση κλπ. Και, τις, και τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Είναι ένα σύνταγμα το οποίο υλοποιείται με νομοθετικά κείμενα μέρα με τη μέρα. Ε, ξεκινήσαμε από τις ε, τοπικές ε, και μάλλον το επόμενο ραντεβού είναι η επόμενη Κυριακή. Έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Για πρώτη φορά θα ψηφίσουν και οι δυνάμεις ασφαλείας. Το Κοινοβούλιο για πρώτη φορά αποφάσισε να τους δώσει το δικαίωμα να ψηφίσουν. Στις 6 Μαΐου θα λάβουν χώρα λοιπόν οι αυτοδιοικητικές εκλογές που θα σηματοδοτήσουν την, το την αρχή της αποκέντρωσης, ε, την αρχή της διαδικασίας αποκέντρωσης. Ε, το Σύνταγμα ήδη μιλάει για ένα αποκεντρωμένο κράτος και οι αυτοδιοικητικές εκλογές αποτελούν την αφετηρία, ε, το πρώτο λάκτισμα αν θέλετε, για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση της αποκέντρωσης η οποία θα αποτελέσει και τη Λιβία Λίθο για το πώς θα γίνει η ανάπτυξη που θα επιτευχθεί η ανάπτυξη στο μέλλον. Ή μην ξεχνάμε ότι η επανάσταση ξεκίνησε από την, το εσωτερικό της χώρας από υποβαθμισμένες περιοχές εξαιτίας τη, του, της διαφοράς που υπάρχει στην οικονομική ανάπτυξη μεταξύ ε, ακτογραμμής των, των παράλληλων περιοχών και του εσωτερικού της χώρας. Οπότε είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ε, εκλογές της 6ης Μαΐου είναι πολύ σημαντικές ε, για τις τοπικές κοινότητες. Αυτή τη στιγμή στην Τινησία υπάρχει εκλεγμένη βουλή, έχουμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας που είναι ερετός. Για πρώτη φορά όμως γίνονται εκλογές σε τοπικό επίπεδο. Ε, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ε, με ένα ακόμα επίπεδο τοπικής διοίκησης ε, σε ε, δήμους και επαρχίες ή περιφέρειες αν θέλετε όπως το προβλέπει το Σύνταγμά μας. Υπάρχει όμως και, άλλο ένα διακύβευμα, είναι η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία. Ο εκλογικός νόμος υποχρεώνει την οριζόντια και την κατακόρυφη ίση συμμετοχή. Ε, δεν θέλουμε απλώς να συμμετάσχουν οι γυναίκες ψηφίζοντας, αλλά και να έχουν παρουσία στα δημοτικά συμβούλια. Τα κόμματα είναι ε, υποχρεωμένα τις εκλογικές τους λίστες να ε, έχουν ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών, αλλά και μεταξύ των εκλεγμένων τους μελών Επίσης, ε, είναι μια προσπάθεια επιβολής της ισότητας, την οποία την ακολουθούμε εδώ και καιρό. Ε, έχουμε ένα πολύ προσφατονομαστικό κείμενο το οποίο αφορά την ασφάλεια των γυναικών και την αποφυγή της βίας εναντίον τους. Επίση και οι νέοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, η συμμετοχή των νέων είναι πολύ σημαντική. Μιλώ για του νέου και τι γυναίκε γιατί θέλουμε να του εμπλέξουμε. Ε, είναι πολύ δυναμικές ομάδες της κοινωνία των πολιτών μα. Ε, είναι ομάδες οι οποίες κατά τη διάρκεια των δύσκολων φάσεων της επανάστασής μας στήριξαν την επανάσταση. Άλλες χώρες δεν είχαν αυτή την ε, ευκαιρία, τη χαρά, την... το προνόμιο. Οπότε σημαντικό διακύβευμα είναι η υψηλή συμμετοχή των, της κοινωνίας, η διοργάνωση των εκλογών είναι πάρα πολύ περίπλοκη, πολύ πιο περίπλοκη από αυτή των κοινοβουλευτικών εκλογών του 2014. Έχουμε πολύ περισσότερους υποψηφίους, για παράδειγμα. Χρειάστηκε σε εισαγωγικά να αποκεντρώσουμε και τα διοικητικά δικαστήρια προκειμένου να στηρίξουμε την, ε, τις τοπικές εκλογές επιτόπου και από το 2011 οι εκλογές στην Τινησία διοργανώνονται από μια ανεξάρτητη αρχή και όχι από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως συνέβαινε κατά την περίοδο της δικτατορίας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντική αυτή η πολιτική στιγμή που θα ζήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Το Συμβούλιο των ε, τοπικών αρχών που θα δημιουργηθεί ε, αμέσως μετά θα δώσει μια πολύ μεγαλύτερη ορατότητα σε αυτή τη διαδικασία. Η την Ισία επίσης δημιούργησε και ένα ανώτατο Συμβούλιο Δικαστικών επίσης πολύ σημαντικό βήμα για την κατοχήρωση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος Αναθεωρούμε συνεχώς την ομοθεσία μας. Το συνταγματικό δικαστήριο επίσης το... αλλάζουμε το νόμο για να, ε, για να δημιουργηθεί ένα συνταγματικό δικαστήριο όπως ακριβώς προλείπει το Σύνταγμα. Θα έχει γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Σε ό,τι αφορά την, την ε, Επιτροπή Αλήθειας και Αξιοπρέπειας, ε, Είμαστε πεπισμένοι για την ε, σημασία μιας ε, ενδιάμεσης προσωρινής δικαιοσύνης. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε πολύ πρόσφατα να σταματήσουν οι εργασίες αυτής της Επιτροπής αλήθειας και της ε, αξιοπρέπειας. Αυτό όμως δεν σημαίνει και το τέλος της ενδιάμεσης δικαιοσύνης, μεταβατικής δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το πώς θα συνεχιστεί. Τα τελευταία 7 χρόνια έγιναν πολλά ολισθήματα. Ο συντονισμός δεν είχε γίνει σωστά. Τώρα προσπαθούμε να συντονίσουμε αυτή τη δράση η οποία θα στηρίξει τη μεταβατική δικαιοσύνη που θα οδηγήσει ε, σε ειρήνευση, σε συμφιλίωση της θυνησίας με το παρελθόν της των τινήσεων μεταξύ τους. Στι 31 Μαου λοιπόν σταματούν οι εργασίε τη Επιτροπή Αλήθεια και Αξιοπρέπεια. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι, ότι σταματά και η δράση τη μεταβατική δικαιοσύνη στην τη δικαιοσύνη τη μετάβαση, δηλαδή, ε, έτσι την ονομάζουμε εμεί, ε, στην Τινησία. Πιστεύουμε ότι η Τινησία συνολικά έχει πετύχει στην δημοκρατική της μετάβαση. Οι ελευθερίες είναι κατοχυρωμένες, πάντοτε και συνεχώς τροποποιούμε κείμενα, ανανεώνουμε την ομοθεσία μας. Ο πρόεδρος ε, ανέλαβε τον περασμένο μήνα, τον περασμένο χρόνο, ε, ανέλαβε μια πρωτοβουλία για την ισότητα ανδρών και γυναικών σε θέματα ε, κληρονομιάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί γνωρίζετε τι προβλέπει ο Ισλαμικός νόμος κλπ. Είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό για μας. Ε, το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πραγματική ελευθερία στην Τινησία, ελευθερία στον τύπο, ελευθερία στα οπτικοακουστικά μέσα, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης η οποία ε, κατοχυρώνεται μέρα με τη μέρα, όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Ζούσαμε για 50 περίπου χρόνια ε, υπό το καθεστώς μιας κατά βάση δικτατορίας. Με ε, ένα μόνο κόμμα, μονοκομματισμό, μία, πραγμα... μία μόνο αλήθεια. Αυτό που έχει συμβεί στην Τινησία είναι μια πραγματική τινησια ειναι μια πραγματικη αλλαγη σε 6-7 χρόνια μετά την Επανάσταση. Δεν είναι και πολλά, σκεφτούμε ότι η χώρα έχει μια ιστορία 3.000 ετών. Σε ό,τι διαφορά την οικονομική μετάβαση, αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες μετά την Επανάσταση, ακριβώς διότι εστιάζαμε στην ε, δημιουργία δημοκρατικών θεσμών. Η δημοκρατία έχει σημαντικό κόστος και το κόστος ήταν οικονομικό. Αν και προχωρήσαμε πάρα πολύ στο πολιτικό επίπεδο, ε, προχωρήσαμε πολύ και στο ε, οικονομικό επίπεδο. Ε, ελευθερία, αξιοπρέπεια και απασχόληση είναι οι τρεις βασικοί μας πυλώνες. Αυτή τη στιγμή η ανεργία είναι στο 15%. πάνω από το 1 τρίτο αυτών είναι απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης και στελέχη. Μετά την Επανάσταση του 2011 η οικονομία ε, ε, ε, άρχισε να ε, μένει πίσω, έμεινε πίσω. Τώρα έχουμε και άλλο ένα θέμα, το θέμα της ασφάλειας, η, την Ισία ως νέα δημοκρατία, καινούργια δημοκρατία, χτυπήθηκε από τρία τρομοκρατικά χτυπήματα το 2015 που, που επηρέασαν πολύ την τουριστική μας κίνηση. Ξέρετε ότι είμαστε η τουριστική χώρα. Όλα αυτά είχαν προγραμματιστεί βέβαια, διότι το κοινωνικό μοντέλο το οποίο αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή δεν συνάδει με το μοντέλο αυτών των τρομοκρατικών ομάδων, Ισλαμικό κράτος κλπ. που μας επιτέθηκαν. και η ασφάλεια στη γειτονιά μας επίσης επηρέασε τις εξέλιξεις μας. Για παράδειγμα η Λιβύη. Το 2011 όταν γινόταν ο πόλεμος στην Λιβύη ε, πάνω από ένα, 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Λιβύη έφτασαν σε μας. Οπότε η κατάσταση της Λιβύης επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και εμάς. Και η τρομοκρατικές δράσεις του 2015 ε, προφανώς ξέρουμε ότι έγιναν από την Ίσιους, αλλά που είχαν συνδέσεις με τη Λιβύη. Η κατάσταση στη Λιβύη μας ανησυχεί ιδιαίτερα και από πλευράς ασφάλειας και από πλευράς οικονομίας, διότι έχουμε πάρα πολύ στενέ σχέσεις με την Λιβύη. Προσπαθούμε να, ε, θα θέλαμε να αναζητηθούν ε, ειρηνικές και διπλωματικές λύσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας ε, ανέλαβε πρωτοβουλίες για να βγει η χώρα από την ε, κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η Τινησία είναι η χώρα η οποία πιο πολύ επηρεάζεται από το πρόβλημα της Λιβύης στην περιοχή μας. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, αυτό είναι το διακύβευμα αυτή τη στιγμή, προκειμένου να πετύχει οριστικά ε, η δημοκρατική μετάβαση. Ε, όπως σας είπα σε πολιτικό πεδίο κάναμε πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την οικονομία αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ανάκαμψη ο τουρισμός ε, ενισχύεται μετά την άρση των περιορισμών που είχε προκαλέσει η ανασφάλεια οι τουρίστες επιστρέφουν. Επενδύσαμε πολύ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στη φυλάξη των συνόρων. Είμαστε πρωτοπόροι στην ε, αντιμετώπιση τρομοκρατίας και μάλιστα έχουμε αναπτύξει και ε, μια ε, τεχνογνωσία πολύ σημαντική. Κανένας βέβαια δεν είναι απόλυτα προστατευμένος. Το είδαμε αυτό ε, και στο Παρίσι και αλλού. Από το 2015 όμως ευτυχώς ε, έχουμε αναπτύξει ένα ε, δίχτυ προστασίας που μας επέτρεψε να μην έχουμε τρομοκρατικά χτυπήματα τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν υπάρχει πλήρης απάλληψη του κινδύνου βέβαια. Οι απειλές υφίστανται. Οι foreign fighters, οι, οι μαχητές, ε, ε, ξένοι μαχητές επιστρέφουν συχνά. Έχουμε ένα, ένα δικαστικό σύστημα το οποίο μας επιτρέπει να χειριστούμε το θέμα. Το 2013 ε, ψηφίσαμε ένα νόμο που έδωσε το, την νομική βάση για θέματα ε, ε τρομοκρατίας και ε, ξεπλήματος χρημάτων ε, που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα θέματα ασφάλειας. Επανερχόμαστε λοιπόν, ανακάμπτουμε οικονομικά, ανταγωνιστικά με τον τουρισμό, με τη γεωργία. Έχουμε αύξηση ε, του 3% το 2018, τουλάχιστον αυτό προβλέπουμε. Ε, για πρώτη φορά τα ε, χρόνια μετά την Επανάσταση. Η μαύρη λίστα ε, μας δημιουργεί προβλήματα. ο κατάλογος Γκάφη, ο κατάλογος ε, ε, του διοντολογικού κώδικα μας δημιουργούν προβλήματα. Προσπαθούμε να βγούμε. Μέχρι το τέλος του χρόνου ελπίζουμε ότι θα έχουμε βγει από τη λίστα Γκάφη σε ό,τι αφορά τον, κατά, τον κατάλογο για την για ε, τον κώδικα διοντολογία. Δεν είμαστε πια στη μαύρη λίστα, είμαστε στην κρύη. Ελπίζουμε θα βγούμε και από εκεί μέχρι το τέλο του χρόνου. Ε, το, τα θέματα αυτά δημιουργούν πολλές ε, φορές δυσκολίες στην κατανόηση. Ε, είναι δύσκολα κατανοούνται από τους πολίτες μας ενώ γιατί θεωρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως στρατηγικό μας εταίρο. Σε ό,τι διαφορά την στρατηγική εταιρική σχέση έχουμε ένα έγγραφο προτεραιοτήτων για το 2018-2019 και σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά το 2020. Θεωρούμε ότι η Τινησία είναι δημοκρατική χώρα. Ε, πριν από την Επανάσταση η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κατηγόρησε πολύ συχνά για θέματα πολιτικά καθεστώτος. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια δημοκρατία, οπότε ζητούμε μια πιο προνομιακή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ε, στενή, ίσως θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ειδικό καθεστώς για την νησία. Ε, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, στις μελλοντικές μας σχέσεις την συμμετρία, ε, την αμοιβαιότητα δηλαδή, και την, το σταδιακό χαρακτήρα. Ε, όπως σας είπα για την τρομοκρατία έχουμε σημαντική τεχνογνωσία. Είμαστε ανοιχτοί σε μια πιο στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή τη στιγμή οι ανταλλαγές ε, υπάρχουν, ανταλλαγές πληροφοριών κλπ, αλλά μπορούν να βελτιωθούν. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι το Open Sky, η ανοιχτή ουρανή. Κάναμε προσπάθειες να υπογράψουμε συμφωνία Open Sky. Αυτή τη στιγμή το μπαλάκι βρίσκεται νομίζω στη δική σας πλευρά, στην πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω ότι υφίστανται ανησυχίες σε ό,τι αφορά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μνημόνιο. Ε, στις 23 του περασμένου Μαρτίου η έκθεση ήταν θετική. Μια επόμενη έκθεση προβλέπεται για τον Ιούνιο. Ε, και έχουμε αναλάβει δεσμεύσει τις οποίες θα, θα υλοποιήσουμε. Ε, Τρία-τέσσερα ακόμα να υπάρχουν, για παράδειγμα κοινωνική ασφάλιση, ε, κρατικές επιχειρήσεις, ε, η κρατική διοίκηση και τέταρτη μεταρρύθμιση που είναι το Ταμείο Αντιστάθμισης ή Αποζημίωσης. Ή το μνημόνιο αυτό μας πιέζει προφανώς, αλλά τις δεσμεύσεις έχουμε αναλάβει και θα τις υλοποιήσουμε. Δεν θα πρέπει οι περιορισμοί που θέτει το Διεθνές Ζωνοτικό Ταμείο να επιβραδύνει την ανάπτυξή μας όμως. Πάντοτε ζητούμε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ε, ενώπιον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Γιατί είμαστε μια νέα καινούρια δημοκρατία. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία τα οποία ήθελα εγώ να υπογραμμίσω. Η Τινησία ε, είναι προσιλωμένη στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Το ε, η ανοιχτή ουρανή είναι ένα εργαλείο συνεργασίας και έχουμε πολλά άλλα τέτοια. Ε, σε ό,τι ε, αφορά όμως την, τον, το προφίλ το, στα, στα μέσα ενημέρωσης το, ε, ε, της σχέσης μας αυτής νομίζω ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί να, γίνει πιο, να γίνουν πιο ορατά τα επιτεύγματα αυτής της σχέσης αυτή τη στιγμή ε, συμμεριζόμαστε τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολίτες μας ε, τις ε, έχουν δεχτεί. Δεν είναι δυνατόν να γίνει υποχώρηση εναντί αυτών. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να δεχτούμε, δεν ποτέ να δεχτούμε την επιστροφή στη δημοκρατία. Θα πρέπει να μετρήσετε σωστά, να σταθμίσετε σωστά το εύρος, των βεληνικές των μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει στην Τινησία. Ε, μετά το δεσποτικό ή δικτατορικό αν θέλετε χαρακτήρα του προηγούμενου καθεστώτος η ε, την εκπέμπει πλέον μια, ένα τελείως καινούριο προφίλ μια τελείως καινούρια εικόνα της ε, δημοκρατίας η δημοκρατία στην Τινησία υπάρχει αναπτύσσεται καθημερινά οι επόμενες ε, επικείμενες ε, αυτοδιοικητικές εκλογές θα την καθιερώσουν ακόμα περισσότερο και θα την ενισχύσουν, θα την εδραιώσουν. Θα πρέπει να βοηθηθεί και ιδιαίτερως ε, στην οικονομική της μετάβαση. Οι Ευρωπαίοι πάντοτε ήταν φίλοι μας και παρόντες για να μας βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας. Τώρα θα περάσουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων, αν συμφωνείτε κι εσείς. Θα δώσουμε το λόγο πρώτα στους συνάδελφους και μετά θα απαντήσουμε ώστε να κάνουμε μια συζήτηση. αν ζω για το ΕΛΚ πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι πρέπει να είστε βέβαιος για το ενδιαφέρον της συνέλευσής μας για την Ισία Τακτικά δείχνουμε ενδιαφέρον για τη μετάβαση στην χώρα σας. Καμιά φορά υπάρχει πίεση να δώσουμε ως παράδειγμα την, ε, την Ισία και νομίζω ότι καμιά φορά αυτή η πίεση είναι υπερβολική ώστε να κάνουμε την Τινησία πρότυπο και μοντέλο για όλη την ε, περιοχή. Οπότε το έργο σας είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια αυτής της ε, μετάβασης. Θα ήθελα, πέρα από τα οικονομικά, να μιλήσουμε λίγο για τα θέματα ασφάλειας. Θα μπορούσαμε βεβαίως να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις, στον είπατε ο ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και κάποιες ε, μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας. Υπάρχει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα της Ένωσης. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα αυτή η διαδικασία. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο από αυτού. Γιατί από ό,τι κατάλαβα αυτή η σχέση αμυνάς και ασφάλειας είναι σε διμερές επίπεδο μεταξύ χωρών της Ένωσης και την Ισίας. Ίσως όχι αποκλειστικά, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς τι γίνεται με αυτή την ε, πτυχή. Δεύτερο ζήτημα. Αναφερθήκατε και εσείς το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εμείς στην Ευρώπη στους ε, επιστρέφοντες μαχητές. Ξέρω ότι υπήρχε ένα σώμα τυνησίων που είχε πολύ ενεργό ρόλο μαχητών Έχετε λοιπόν κάποια άλλα στοιχεία σε σχέση με την ε, επάνωδο αυτών των μαχητών ή την ε, παρουσία, παρουσία τους σε άλλα θέατρα πολεμικά της Τσιχάντ. Ευχαριστώ τον κύριο Ταζάν. Θέλετε να απαντήσετε μία-μία τις ερωτήσεις ή ανομάδες. Ωραία, ανομάδες ερωτήσεων. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Βερσιάκη μέρους της ΓΚΟΕ. Καλημέρα κύριε Πρωθυπουργέ. Εδώ είμαι. Αν δεν με βλέπετε, εδώ είμαι. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ στην Επιτροπή μας. Λυπάμαι που τον περασμένο μήνα δεν μπορέσαμε να συναντηθούμε στην την Ισία και λυπάμαι γι' αυτό και στο συγγνώμη εγώ. Είναι σημαντικό αυτό που είπατε, ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να συνοδεύουμε την Τινησία προς την δημοκρατική μετάβαση. Εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε. Παρόλο που δεν θα έχουμε αποστολή παρατηρητών για τις τοπικές εκλογές, θα παραβρεθούμε, θα έρθει και ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Καστάλντο, για τις τοπικές εκλογές θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι αρμοδιότητε των ε, οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης που θα προκύψουν πρώτα αυτό. Δεύτερο, για αυτή τη μαύρη λίστα της τρομοκρατίας την οποία αναφέρατε αρχίζουμε να βλέπουμε να ελοποιούνται κάποιες ε, υποσχέσεις σε αυτό το θέμα. Το ΑΛΕΚΑ η Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών. Ίσως θα ήταν προτιμητέο να είχαμε μια συμφωνία εταιρική σχέση, όχι μόνο ελευθερών συναλλαγών. Οπότε θα πρέπει εμείς να τονίσουμε τη σημασία αυτής της συμφωνίας και τον κίνδυνο για την γεωργία στην Τινησία. Οπότε τι γίνεται και με αυτό το θέμα, θα ήθελα να μου το αναφέρετε. Τι γίνεται επίσης με το ελαιόλαδο και κάτι άλλο. συναντήθηκα με αλληλείς από το Ζαρζής την περασμένη εβδομάδα ε, που ανησυχούν κάποιες ποσοστώσει όσον αφορά την αλία του τόνου. Θα ήθελα να μου πείτε κάτι και γι' αυτό και για την κινητικότητα επίσης. Θεωρείτε ότι οι τωρινέ διαπραγματεύσει επιτρέπουν μία ισοβαρή διαπραγμάτευση και όχι μόνο μονομερή, δηλαδή επανασδοχή των υπηκών τρίτων χωρών που διέρχονται από την, ε, Ισία και λύγεται με τι θεωρήσεις. Και κάτι άλλο επίση να αναφέρω, αναφερθήκατε στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πράγματι υπάρχουν αναφεσβήτητε πρόοδοι, υπάρχουν όμω δύο ζητήματα τα οποία παραμένουν και τα οποία καταγγέλλονται. Οι βασανισμοί, τα βασανιστήρια, η αστυνομική αυθαιρεσία Ξέρετε ότι αυτό το έχουμε συζητήσει επανειλημμένω και θα ήθελα να μου δώσετε κάποιες εξηγήσει σε σχέση με την Επιτροπή αυτή αληθεία και αξιοπρέπειας ή συμφιλίωσης. Διορθώνει η μιλήτρια τώρα, τωρα αληθεια και αξιοπρέπειας. Γιατί υπάρχει μια πολεμική γύρω από αυτή την Επιτροπή. Θα ήθελα τα σχόλιά σα και σταματάω εδώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. ο κ. Γιούρα και Παρακαλώ, συνάδελφοι, να τηρήσετε τη χρονομιλία σα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Πρωθυπουργό για τι ε, πληροφορίε του. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Η Τινησία είναι εγγύης χώρα στην Ευρώπη και πολιτικά και γεωγραφικά. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, ενημερωθήκαμε για μία αύξηση της παράνομης μετανάστευσης από την Τινησία. Παρόμοια μετανάστευση που αφορά την ίσιους υπηκόους. Πώς ερμηνεύετε εσείς αυτό το φαινόμενο αύξησης μετανάστευσης των δικών σας πολιτών. Δεύτερον, έχουμε κάποιες ε, πληροφορίες από κάποιες οργανώσεις όσον αφορά διακριτική μεταχείριση χριστιανών. Τι γίνεται με τις νομικές διακρίσεις ε, και την ε, καταπίεση αυτών των ανθρώπων. Προστατεύονται αυτοί οι χριστιανοί οι οποίοι έχουν αλλαξοπιστήσει από την Τινησία, από τις Τινησιακές Αρχές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Γιούρεκ, ο κύριος Μαρσελεζή για τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να σας πω καταρχάς ότι η Τινησία για μας δεν είναι μόνο ένας γείτονας, αλλά κυρίως ένας σύμμαχος, ιδιαίτερα στην τωρινή κατάσταση όπου είναι η μόνη χώρα στο Μαγκρέπ που πιστεύουμε ότι είναι η μόνη που πηγαίνει προς την δημοκρατία. Και αυτό ακριβώς μας εκπλήσει που καμιά φορά βλέπουμε ότι κάποια τμήματα της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μεταχειρίζονται την, την ΣΥΑ ως ένα παραπάνω γείτονα αντί ως ένα σύμμαχο. Είμαι Ισπανό, ξέρω πόσο καιρό χρειάζεται η μετάβαση στη δημοκρατία, δεν τελειώνει σχεδόν ποτέ, είναι μια εξελεκτική διαδικασία και θα σας στηρίξουμε απόλυτα σε αυτή τη διαδικασία. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Άκουσα αυτό που, που είπατε για τη μεταβατική φάση της δικαιοσύνης. Έχω κάποιες ανησυχίες και θα ήθελα να μάθω τα εξή. Τι γίνεται με τις διώξεις σε σχέση με τους συνεργάτες του καθεστώτος Μπεναλή και το δικαίωμα των θυμάτων για αποζημίωση. Τώρα για την ΑΛΕΚΑ συμφωνώ απόλυτα. Θα πρέπει να υπάρχει συμμετρία, θα πρέπει να υπάρχει εξελικτικός χαρακτήρας και θα ήθελα να μου πείτε αυτό το είδος εμπορική συμφωνίας θα μπορούσε να συνδεθεί με την κλιματική συμφωνία του Παρισιού και την ε, βιώσιμη ανάπτυξη γιατί νομίζω ότι αυτό θα αποτελούσε ένα πολύ καλό τρόπος να καταλήξουμε συμφωνίε εμπορικέ, οι οποίε ήταν βιώσιμες και θετικέ για όλου. Επίση για το ενεργειακά σα συστήματα, δεν ξέρω αν το αναφέρατε αυτό, για τα διάφορε μελέτε για την, ε, την έχουμε και την συμφωνία του Παρισιού. Μήπως έχετε ξεκινήσει η διαδικασία από ανθρακοποίηση στην ε, νησία και ποια είναι η προθεσμία, το χρονοδιαγράμμα σα. Και άλλο ένα ζήτημα, όχι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό, τι γίνεται με τα νητρόδη, ε, τι γίνεται με τα επίπεδα καρμίου τα οποία είναι αποδεκτά. Ε, θα θέλαμε να υπάρχουν χαμηλότερα επίπεδα ώστε ακριβώς να προστατεύεται η υγεία και το περιβάλλον και τι χρειάζεται να κάνουμε εδώ ώστε να βοηθήσουμε τη βιομηχανία σας για να ανταποκριθεί ακριβώς στις προδιαγραφές υγείας και ε, περιβάλλοντος που έχουμε στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστούμε. Τρεις τελευταίοι ομιλητές. Ο κύριος Καστάλτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Με χαρά και με τιμή σας ε, υποδεχόμαστε σήμερα στην Επιτροπή μας των Εξωτερικών Υπαθέσεων Επανειλημμένως στην ευκαιρία να υπογραμμίσω το στρατηγικό ρόλο της Τινησίας στην περιοχή, στη Μεσόγειο γενικότερα, ως εισηγητής παλαιότερα στο Κοινοβούλιο εδώ. Και βεβαίως χαιρετίζω με μεγάλη χαρά τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις για τη νομοθετική εργασία που προτίθεστε να κάνετε το τελευταίο διάστημα και το οποίο υπογραμμίσατε. Ε, Βεβαίω έχω και την τιμή να ηγούμε αυτή της αποστολής παρατηρητών που θα λάβει η χώρα την ερχόμενη εβδομάδα για τις τοπικές εκλογές. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω κάποιες ερωτήσεις από αυτού γιατί ξέρω ότι στο παρελθόν, ιδιαίτερα πέρσι, είχαμε κάποια μπλοκαρίσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανεξάρτητη αρχή για τις εκλογές. Ο πρόεδρος της είχε παρετηθεί μετά από έντονες επικρίσεις. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν το κλίμα έχει βελτιωθεί. και αν θα γίνουν όλα τα απαραίτητα ώστε να ξεκινήσουν ομαλά οι εκλογές. Επίσης να ρωτήσω ποιες είναι οι πολιτικές επιπτώσεις που θεωρείται θα έχουν αυτές οι εκλογές σε εθνικό επίπεδο. Ε, ναι, βεβαίω, είναι τοπικές εκλογές, όμως θα δεξαχθούν σε όλους τους Δήμους, σε όλες τις πόλεις της χώρας. Οπότε θα αποτελούσουν μια δοκιμασία για όλα τα πολιτικά κόμματα που θα έχουν αντίκτυπο παντινησιακό Επίσης, άλλη μία ερώτηση για τη Λιβύη. Είδαμε κατά διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης τη δέσμευση της χώρας, σας, της χώρας σε πολιτικό και δικαστικό επίπεδο ώστε να υπάρξει πραγματικά οικονομική και κοινωνική πρόοδος. Αλλά στη Λιβύη, ας πούμε, έχουμε το θέμα της υγείας του κυρίου Αφτάρ. Οπότε, εδώ τι επίπτωση έχει αυτό το ζήτημα στη χώρα σας του ισχυρού ανδρός της Κυριναϊκής. Τι γίνεται με τον έλεγχο των συνόρων, γιατί ξέρω ότι έχετε κάνει κάποια σημαντικά πράγματα όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων. Και για το θέμα της μαύρης λίστας. Εμείς ελπίζουμε σύντομα να τηρηθούν αυτά που έχετε υποσχεθεί, υποσχεθεί ώστε να προχωρήσετε. Επίσης, τι γίνεται με την ε, συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τα ποσοστά υποψηφίων νέων και γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Καστάλλο και ο πρόεδρος, ο κύριος Μιχαλ Γκάλερ τώρα. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Βάλτε τα ακουστικά σας παρακαλώ. Ωραία, σας καλωσορίζω. Κύριε Πρωθυπουργέ, χαίρομαι που λίγο πριν από τις τοπικές εκλογές βρίσκεστε εδώ. Το κανάλι 3 βάλτε παρακαλώ. Αλλά δεν fängt die Zeit auch nochmal neu an, bitte, ja? Ο χρόνος μηδενίζεται όμως, ε. ξεκινάω από την αρχή, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, τα ξαναλέω λοιπόν. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ λίγο πριν ε, τις ε, τοπικές εκλογές που θα γίνουν στην Τινησία. Εγώ ήμουν επικεφαλής των παρατηρητών το 2011 ε, για τη συντακτική συνέλευση και χαίρομαι πολύ που επιτέλους διοργανώνονται αυτές τις τοπικές εκλογές με μια μικρή καθυστέρηση βέβαια πρέπει να πούμε και Χαίρομαι μάλιστα ότι ε, μία από τις συστάσεις του 2011 ήταν ε, και η συμμετοχή και των ενόπλων δυνάμεων, των ε, μελών των ενόπλων δυνάμεων στην εκλογική διαδικασία. Αυτό θα γίνει τελικά και θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε η συνάδελφος Βερζιά. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης και ποια θα είναι η χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, αυτή η νέα μορφή δημοκρατικής νομιμοποίησης θα μπορούσε να συμβάλλει στην εγγέννη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας. Ε, θεωρώ ότι ένα από τα προβλήματα της Τινησίας σχετίζονται με το γεγονός ότι η κεντρική κυβέρνηση είναι υπερβολικά συγκεντρωτική. Ίσως λοιπόν η ε, απονομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε χαμηλότερο επίπεδο, στο τοπικό και περιφερειακό, θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίλυση των ε, προβλημάτων της χώρας. Ε, γιατί ακριβώς ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο να αρθούν και προβλήματα που σχετίζονται με δυσκινησία, δυσλειτουργία ή και διαφθορά ακόμη. Για το κληρονομικό δίκαιο Αναφερθήκατε στο, στην ομιλία του Προέδρου. Ποια θα είναι τελικά η κατάληξη αυτής της διαδικασίας. Οι άνδρες και οι γυναίκες θα έχουν ίσα δικαιώματα στο κληρονομικό δίκαιο. Θα καταλήξουμε σε μια μεικτή μορφή δικαίου, όπου ενδεχομένως θα είναι προαιρετικό, να μπορεί δηλαδή μια γυναίκα ε, να έχει δικαίωμα ε, κληρονομιάς. Ε, επίσης, ε, Αναφερθήκατε στην επιστροφή στη χώρα σας ξένων μαχητών. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε πρόβλημα και με την ίσιους υπηκόους και την επανεισδοχή τους, ε, την επιστροφή τους στη χώρα. Γιατί ε, τέθηκαν και διάφορα διαδικαστικά θέματα και στη Γερμανία. Ε, έχουν λυθεί πλέον αυτά τα διαδικαστικά θέματα στη χώρα σας, μπορούν να επιστρεφούν οι άνθρωποι αυτοί. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Είπατε ότι η κατάσταση στον τουρισμό ε, βελτιώνεται. Μπορείτε να μας δώσετε συγκεκριμένους αριθμούς, στοιχεία. Έτος αναφοράς προφανώς είναι το 2010. Ε, ελπίζω να βελτιωθεί και εγώ η κατάσταση στον τουρισμό, να έρθουν πολλοί Ευρωπαίοι στη χώρα σας για να συμβάλλουν και αυτοί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας σας. Ευχαριστώ. Κύριος καλώς ήρθατε θα ήθελα να ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένος. Είχατε ήδη ξεκινήσει την παρέμβασή σας. Ε, πάση περιπτώσει, ερχόμουν από την Επιτροπή Αλίας. Ξέρω ότι ήσασταν υπουργό Αλίας παλιότερα, οπότε παρακαλώ πολύ επίοικια. Ε, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής ε, ε, στη δημοκρατική πρόοδο που έχετε καταγράψει. Ε, και στην αντιμετώπιση της ε, τρομοκρατίας. Είστε μια δημοκρατία μοντέλο για άλλες χώρες πλέον. Και σας καλωσορίζω θερμά. Θα ήθελα να μου πείτε δύο, δύο λόγια περισσότερα για το ποιο πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ακριβώ το καθεστώ των σχέσεων μεταξύ τη Ισία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή έχετε, ε, είσαστε στην ανώτερη ταχύτητα του καθεστώτος εταιρική σχέση. Ε, τι όμω ακριβώ έχετε στο μυαλό σα. Ε, ο, την περασμένη ομιλία ε, συστήσαμε, ε, υιοθετήσαμε ένα κείμενο και ο κ. Χάν είχε πει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το ε, εργαλείο της γειτονίας στην οικονομική μας στρατηγική του 2020. Ε, ποια είναι η δική σας άποψη ακριβώς. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε, όπως συζήτησε ο κ. Γκάλερ, να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για τον τουρισμό και για τις εξωτερικές επενδύσεις. Λέτε ότι η απασχόληση είναι μία από τις σημαίες της επανάστασης στην Τινησία. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε για το σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι εξωτερικές επενδύσεις. Τέλος, ε, ο, αριθμητικά στοιχεία για την ε, μετανάστευση από την Τινησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχετε προβλήματα με λάθρο μετανάστευση ε, και ε, το πώς πιστεύετε ότι πρέπει να διευκολυνθούν οι καθηγητέ, οι φοιτητέ κλπ. για να έχουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε συνάδελφοι για τα πολλά αυτά ερωτήματα, τις παρεμβάσεις σας. Κύριε Σάιντ, έχετε 10 με 15 λεπτά περίπου για να απαντήσετε. <laughs> bon. Euh, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και τα ερωτηματικά. Είναι και ευκαιρία για μας να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα που καμιά φορά δεν είναι και τόσο σαφή σε επίπεδο ε. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια ελλείμματα όσον αφορά την ενημέρωση για τα συμβάντα στην Τινησία, κάτι το οποίο θα πρέπει να βελτιώσουμε και να δώσουμε πιο, περισσότερες και σωστότερες πληροφορίες. Διάφορα ζητήματα τέθηκαν. Καταρχάς για την ασφάλεια. Πράγματι έχουμε ένα πρόγραμμα συνεργασίας με την Ένωση. Είναι πιο εύκολο η διμερής συνεργασία για αυτά. Από ότι με την Ένωση είναι αλήθεια αυτό. Αλλά για το πρόγραμμα νομίζω ότι υπήρξε ένα μικρό μπλοκάσμα το οποίο θα ρυθμιστεί, θα λυθεί τις επόμενες μέρες. Τώρα για τις δυνάμεις από την Τινησία που έχουν παρουσία στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στη Λιβύη, εμείς στην Τινησία εντοπίσαμε γύρω στους 3.000 πολίτες της Τινησίας. Αυτά τα στοιχεία δώσαμε εξάλλου και τα ενημερώνουμε καθημερινά. Πολλοί απεβίωσαν, πέθαναν στη μάχη, κάποιοι βρίσκονται στη φυλακή. Έχουμε αποστολές ασφαλείας ε, τακτικές ώστε να ενημερώνουμε συχνά τις λίστες και να δίνουμε περισσότερες πληροφορίες. Ξέρω ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ανησυχούν και μου το εκφράζουν στις συναντήσεις μου οι επικεφαλής των κυβερνήσεων. Εμείς στην Τινησία πέρασαμε ένα νόμο το 2015 κατά της ε, τρομοκρατίας και της ε, νομιμοποίησης προσόδων και η αποστολή Γκάφη που ήρθε στην έλαβε χώρα πριν την, την ε, ψήφιση αυτού του νόμου. Οπότε δεν το έλαβε υπόψη της στην αξιολόγησή της. Πρόλη πάντως αυτός ο νόμος ότι όλοι οι τινήσιοι που έχουν συμμετάσχει σε δράσεις ε, τρομοκρατικές στο εξωτερικό αμέσως συλλαμβάνονται στο, στο αεροδρόμιο. Το μικρό πλαίσιο μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Βέβαια θα πρέπει να προσέχουμε γιατί έχουμε μία επάνωδα αυτό των ξενομαχητών προς τη Λιβύη με αυτά που έγιναν με το ΔΑΕΣ στη Μοσούλη και στην ε, Συρία έχουμε μια ροή ε, συμπληρωματική που αφορά εμάς. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι έχει κέρια σημασία το θέμα της ασφάλειας, ναι. βέβαια, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχα πει ε, μάλιστα παλαιότερα ότι εμεί ως την Ίση, την Ισία προστατεύουμε τα νότια σύνορα της Ευρώπης. Είχαμε επιθέσει στη Λιβύη, και επιθέσεις αλλού όπως το Μάντσεστερ που είχαν προετοιμαστεί στη Λιβύη Οπότε θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί και να ε, παγρυπνούμε. Έχουμε 500 χιλιόμετρα σύνορα με την Λιβύη και προσπαθούμε να τα εξασφαλίσουμε σε συνεργασία με τους φίλους μας τους Γερμανούς ηλεκτρονικά και βέβαια είχαμε ανοιχτά σύνορα λόγω ακριβώς της εγκύτητας με τον ε, λιβικό λαό και των ε, αδελφικών ιστορικών σχεσεών μεταξύ μας. Είναι πάντως ε, πραγματικό πρόβλημα αυτό της επανόδου των μαχητών και προσέχουμε βεβαίω για ενδεχόμενες διεισδύσεις και φιλτραρίσματα. Και εδώ βέβαια αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη τρομοκρατική απειλή. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε μία προσέγγιση γιατί ε, η αποκλειστική προσέγγιση έδειξε τα όρια και τους περιορισμούς της, θα πρέπει να περάσουμε σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση και για την ασφάλεια, αλλά να περιλάβουμε εδώ και την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ώστε να προσπαθήσουμε να προσανατολίσουμε αυτά τα άτομα, να αποφύγουμε την μετάβασή τους στην τρομοκρατία και να καταπολεμήσουμε διεθνώς τον εξτρεμισμό και την τρομοκρατία σε συνεργασία με πολλές χώρες, βασιζόμενοι στην εκπαίδευση, στο πολιτισμό, εστιάζοντας ε, στους νέους, στην νεολαία, η οποία η οποία είναι αυτή που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο μετάβαση προ την παραμετα... μετανάστευση και την τρομοκρατία. Είχαμε περιπτώσει τρομοκρατία στην Ευρώπη που δείχνουν ότι σήμερα η απειλή βρίσκεται παντού Έχουμε και το έγκλημα στον ε, κυβερνοχώρο. Ο Τινίσιος που έκανε την ε, τρομοκρατική ενέργεια στη Γερμανία έφυγε από την, την ισχύα του 11. Τότε δεν είχαμε καμιά ένδειξη ότι ήταν τρομοκράτης. Ήταν ένας παράνομος τότε, αλλά δεν ήταν τρομοκράτης. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είναι πολύ σημαντική η συνεργασία στα θέματα της ασφάλειας. Είναι μια παγκόσμια απειλή που αντιμετωπίζουμε εξελίσσεται παντού σε όλη την φίλη. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας και τους δεσμούς μας όσον αφορά την ασφάλεια και την ανταλλαγή πληροφοριών. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που αναφέρθηκε, οι τοπικές εκλογές. Οι δημοτικές αυτές εκλογές ήταν μια μακροχρόνια διαδικασία και για να καταλήξουμε εκεί εφαρμόσαμε τρία κυρία στοιχεία την ε, διοικητική χωροτακτική κατανομή ώστε να καλύπτεται το σύλλογο της επικράτειας και όλοι να έχουν υπηρεσίες δημοτικές και πρόσβαση. Γι' αυτό ακριβώς κάναμε μια κατανομή ώστε να έχουν όλοι πρόσβαση. Δεύτερον, φλογικός νόμος που όπως είπα μας επιτρέπουν να έχουμε ψηλό αριθμό γυναικών και νέων και ατόμων με μειωμένη κοινικότητα επίσης, γιατί το περιλάβαμε στην νομοθεσία. Μετά, ο κώδικας για τις συλλογικότητες που θα συζητήσουμε τώρα, που θα θεσπίσει ακριβώς τα δικαιώματα σε περιφερειακό επίπεδο. Επειδή σήμερα συζητάμε στην χώρα τι ακριβώς ε, δικαιοδοσίες θα έχουν οι περιφέρειες, τι γίνεται με τους δημόσιους υπαλλήλους στις περιφέρειες γιατί οι δύο κύριες προκλήσεις για την επιτυχία της αποκέντρωσης είναι ακριβώς η ανθρώπινη πόροι και η οικονομική πόροι βέβαια στις περιφέρειες. Υπάρχει χαμηλό ποσοστό οικονομικής ε, αυτονομίας για αυτές τις περιφέρειες, οπότε αυτό αποτελεί μια πρόκληση για να πετύχουμε τη διαδικασία ακριβώς αποκέντρωσης, διαδικασία που ενδεχομένω να τρομάζει κάποιους, γιατί είχαμε συνηθίσει την κεντρική εξουσία στην κεντρικοποιημένη εξουσία στην ε, την και γι' αυτό ακριβώ ε, προβλέψαμε μια διαδικασία που θα διαρκέσει κάποια χρόνια. Ξέρω βέβαια ότι σε διάφορε χώρε τη Ευρώπη θα δείτε ότι αυτό συνεχίζεται. Θα δείτε, μου έλεγε ένα Βόλγο φίλο, ότι ακόμα και σήμερα στο βιβλικό τύπο γίνονται συζητήσει για την αποκέντρωση. Για το ελαιόλαδο. Εμείς ζητήσαμε μια επιπλέον ποσόστοση από την Ένωση γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό προϊόν για την Τινησία. Εμείς δεν θέλουμε όμως να αποτελέσει ένα είδος παζαριού με τους εταίρους μας της Ένωσης. Κυρία Βερζιά, για την ιστορική σας παρέμβαση στην Τινησία τη γνωρίζουμε όλοι απ' έξω για το ΑΛΕΚΑ, τη Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών. Βρισκόμαστε σε μια φάση δύσκολης ε, οικονομικής μετάβασης. Υπάρχει μια σημαντική πίεση στα δημόσια οικονομικά μετά από αυτά που έγιναν στην Επανάσταση. Η κυβέρνηση που ακολούθησε ε, υποχρέωθηκε να κάνει πολλές προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων. Τώρα ε, έχουμε και προσταξιδοτήσει ακριβώ για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο και μέσω τη ΑΛΕΚΑ βέβαια αυτή τη συμφωνία των θέσεων υπάρχουν κάποιοι φόβοι. Ξεκινήσαμε λοιπόν διάλογο με την κοινωνία των πολιτών για να εξηγήσουμε ότι αυτή η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών αποτελεί μια ευκαιρία για την χώρα αν τη διαχειριστούμε σωστά. Να σε υπόψη ότι είμαστε τελείω διαφορετικέ οικονομίε, οπότε θα πρέπει να προσδοκάμε βεβαίως ένα δικό χάρτη, αλλά με προσήλωση. Γιατί η Ευρώπη είναι σημαντικός μας εταίρος. 75% συναλλαγών μας γίνονται με την Ευρώπη και πολλές επιχειρήσεις τους ε, είναι παρούσες στην ε, χώρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικός εταίρος και αυτή η συμφωνία αποτελεί μια συμφωνία που διευκολύνει το πλαίσιο των ανταλλαγών μεταξύ των δύο. Άλλη ερώτηση. Επιτροπή Αληθείας και Αξιοπρέπειας. Δεν σημαίνει ότι σταματά το έργο της δικαιοσύνης. Είχαμε μια απόφαση από τους εκπροσώπους του λαού, τους βουλευτές δηλαδή που ψήφισαν αυτό το διάταγμα στις 31 του μήνα και κάποιοι βουλευτές από ένα άλλο κόμμα θεώρησαν ότι αυτή η Επιτροπή Αληθείας και Αξιοπρέπειας θα πρέπει να σταματήσει στις 31 Μαΐου. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα σταματήσει βέβαια και το έργο της δικαιοσύνης. Αυτό ψήφισαν αυτοί οι βουλευτές. Ε, δεν το ψήφισαν επειδή θεωρούν ότι έχει απομακρυνθεί από, την, ε, από το έργο της. Σήμερα βρισκόμαστε μια φάση αποζημιώσεων, δημοσίων υπαλλήλων κτλ. Και σήμερα πια θα πρέπει να αναζητήσουμε ένα εργαλείο το οποίο θα πρέπει να μας επιτρέψει να συμφιλιώσουμε τους την με το πρόσφατο παρελθόν και η δικασίες που έχουν ξεκινήσει και συστάσεις ήδη έχουν σταλεί στη δικαιοσύνη για την εξέταση όλων αυτών των υποθέσεων. Κάποια άλλα στοιχεία που θέσατε, τουρισμός. Όπως ξέρετε είχαμε τρεις μεγάλες τρομοκρατικές ενέργειες το 2015 κατά του τουρισμού και μετά άλλαξε η φυσιογνωμία των τουριστών που έρχονται στην Τινησία. και πάνω από δύο εκατομμύρια Αλγερινοί έρχονται στην ε, την νησία. Και έχουμε τον τελευταίο καιρό μετά από εξελίξεις επάνωδο επιστροφή των Ευρωπαίων τουριστών. 7 εκατομμύρια, 3 από την ε, Αλγερία και οι γειτονικέ χώρες, 2 εκατομμύρια Ευρωπαίων, κυρίω Ιταλών και οι προοπτικέ είναι πολύ θετικέ για το 2018. Αναμένουμε 8 εκατομμύρια τουρίστε με πολύ σημαντικό ποσοστό επανόδου Ευρωπαίων τουριστών. Ε, λόγω ακριβώ τη αύξηση του επίπεδου ασφαλεία. Παρόνομη μετανάστευση. Τώρα. Έχουμε την κατάσταση στη Λιβύη. Είχαμε ένα παράτυπο κύμα μετανάστευση αυτού του είδους και προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε. Για την κινητικότητα και τη συνεργασία είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε μορφή συνεργασία, επαναεισδοχή ή ε, αύξηση τη ποσόστοση για του τιμήσιου. Νομίζω πάντω ότι η μετανάστευση των τιμησίων βεβαίω έχει να κάνει με την χώρα προέλευση. Έχουμε βεβαίω και τη μετανάστευση εξειδικευμένων ε, θυμίσιων που πηγαίνουν παντού στην Ευρώπη και που συμβάλλουν επίσης στην ε, επιμερία της χώρας τους. Μετά, για τον άνθρακα, δυστυχώς ε, δεν ξέρω να σας απαντήσω γιατί είναι πολύ περίπλοκο το θέμα για μένα. Η βία από, και η αυθαιρεσία η αστυνομική. Βλέπω ότι και σε εσά τις χώρες σας εδώ της Ευρώπης ε, συμβαίνουν αντίστοιχα φαινόμενα. Έχει ξεκινήσει πάντως έρευνα δικαστική Υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι τιμωρήθηκαν, συνελήθησαν, φυλακίστηκαν και βεβαίως η μεταμόρφωση ενός δικτατορικού κράτους σε μια δημοκρατία είναι κάτι το μακροχρόνιο, είναι κάτι το οποίο είναι μια εξελεκτική μασιακή διαδικασία και σήμερα εκπαιδεύουμε την αστυνομία να γίνει ένα δημοκρατικό όργανο και να αντιμετωπίσει βέβαια διάφορες προκλήσεις όπως εξτρεμισμός, τρομοκρατία, με τις μορφές που την συναντάμε σήμερα και με όλες αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε και να επαγρυπνούμε ώστε ό,τι γίνεται να γίνεται σεβόμενη τον νόμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Πρέπει όμως να κατανοήσετε αυτή την αλλαγή, αυτή τη μεταμόρφωση που ήταν ριζική στην Τινησία. Ε, πολλές χώρες, ε, όπως η Ισπανία, είχαν αντίστοιχε εμπειρίες και εδώ βρισκόμαστε παρά 7 χρόνια μετά την Επανάσταση. Έχουμε χρόνια ιστορία, χιλιάδων χρόνων. Ε, θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε αυτή τη διαδικασία γιατί έχουμε και θέματα ασφάλειας και έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στο σκέλος της ασφάλειας. δεν είχαμε μεγάλε επενδύσει στα θέματα άμυνα, γιατί έχουμε καλέ σχέσει με τι γειτονικέ μα χώρε, αλλά έχουμε αυτή τη νέα πρόκληση της ε, τρομοκρατίας που προσβάλλει τη δημοκρατία. Οπότε α λάβουμε υπόψη μα ότι έχουμε αυτή τη ριζική αλλαγή στο πολίτευμα και βεβαίω ζητάμε τη στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη νέα νεαρή δημοκρατία. Δεν είναι ένα διακύβευμα μόνο δημοκρατικό αλλά στρατηγικό και γεωπολιτικό. Ε, δεν είναι μόνο το θέμα το οικονομικό, αλλά το ότι προσπαθούμε να προσπίσουμε τις ίδιες αξίες που ισχύουν εδώ στην Ευρώπη, γιατί οι νέοι, οι τινήσιοι επαναστάτησαν ακριβώ για να ζήσουν μέσα στην αξιοπρέπεια, όπως ακριβώς στην Ευρώπη. Έχουμε ισχυρή παρουσία της κοινωνίας των πολιτών, έχουμε υψηλό επίπεδο αλφαβητισμού, έχουμε την κατάσταση γυναικών η οποία είναι πολύ καλή, οι γυναίκες είναι ελεύθερες, υπάρχει ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, και μυστολογικά, Βέβαια, εντάξει, θα πρέπει να γίνουν κάποιε προσπάθειες ακόμα και ψηφίσαμε ένα πολύ σημαντικό νόμο που καταπολεμά τη, τη βία κατά των γυναικών. Παραμένουν λοιπόν σημαντικέ προκλήσει αυτή τη στιγμή και θεωρούμε ότι ο κύριος εταίρος μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να μας βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη μεταβατική φάση. Ξέρω ότι ο χρόνος μου περιορίστηκε και θα σταματήσω εδώ. Thank you. Κύριε Τσαέντ, Ευχαριστώ πολύ. Μάλλον δευτερολογήσατε όπως στο Κοινοβούλιο της Τινησίας, αλλά απαντήσατε λεπτομερώς. Να ενημερώσω επίσης ότι η αποστολή της Επιτροπής ΑΦΕΤ ε, θα επισκεφθεί την, ε, την Ισία και την Αλγερία τον Ιούλιο. Ε, δεν έχουμε ακόμα συγκεκριμένε ημερομηνίε. Αν είστε διαθέσιμος όμως, θα ήταν χαρά μας να συνεχίσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχόμαστε μια καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Ταγιάννη σήμερα το απόγευμα και συνέχεια μια ασφαλή μετάβαση στο Λουξεμβούργο και στις κάτω χώρες όπου θα έχετε διμερείς συνομιλίες. Θα θέλαμε να σας ξαναευχαριστήσουμε για το χρόνο που μας αφιερώσατε για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα που αφορούν μια χώρα που γνωρίζετε ότι είναι πολύ σημαντική για μας. Θα θέλαμε να ε, ε, σας ευχαριστήσουμε και για το εξαιρετικό έργο του πρέσβη σας εδώ στις Βρυξέλλες. Είναι πάντοτε χαρά μας να συνεργαζόμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή τύχη. Colleagues. Συναδελφοί, έχουμε αργήσει λίγα λεπτά, οπότε περνάμε στο σημείο 16 της σημερινής ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Νιζάρ Χαϊ Ραλά, αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών του Ιράκ, Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υπερθέσεων. Είναι χαρά και τιμή μας που είστε εδώ. Ο κύριος Χαραλά είναι, ε, η επίσκεψή του γίνεται σωστό ε, χρονικό ε, σημείο. Χθες μόλις έγινε μια πρώτη συζήτηση για την Συμφωνία Συνεργασία και Εταιρική Σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιράκ και γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει το πράσινο φω προτού τεθεί σε πλήρη εφαρμογή και ισχύ η συμφωνία αυτή. Είδαμε πολλά θέματα χτε. Τα πράγματα προχωρούν στο Ιράκ. Πριν από δύο μήνε το Κουβέιτ ε, φιλοξένησε μια συνδιάσκεψη για την ανοικοδόμηση του Ιράκ και στι 12 Μαου θα διεξαχθούν εθνικές εκλογές στη χώρα σας. Θα θέλαμε να μας πείτε τη δική σας άποψη για το πώς προχωρούν τα πράγματα στη χώρα σας. Έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Ιρακινή κυβέρνηση έχει καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να τίνει χείρα συνεργασίας στους γειτονέ τη, και θα θέλαμε να μας πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες του Ιράκ στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και βεβαίως στο περιφερειακό πλαίσιο της ε, περιοχής σας. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω τον λόγο για 10-15 λεπτά και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να σας συναντήσω εδώ στις Βρυξέλλες. Η σχέση ανάμεσα στο Ιράκ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις προτεραιότητές μας ε, στην εξωτερική μας πολιτική. Ε, ε αναζητούμε μια μακρόχρονη, μακροπρόθεσμη συνεργασία. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι το πιο, πιο σημαντική ομάδα χωρών που μπορεί να βοηθήσει το Ιράκ στην μεταπολίτευση του, τη, μετάβαση, τη μετάβασή του στη δημοκρατία. Και προσπαθούμε πάρα πολύ σκληρά να πετύχει αυτή η μακρόπνοη συνεργασία στο Ιράκ έχουμε σημαντικά επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια. Η συνεργασία μας με την Διεθνή Συμμαχία ε, κατόπιν της ανάγκης να καταπολεμήσουμε τον, το Ισλαμικό κράτος κατόπιν αιτήματος του ΟΗΕ ε, δεχτήκαμε στήριξη στρατιωτικού συμβούλους κλπ μαχητές, προσωπικό, στρατιώτες ε, τα καταφέραμε και τώρα θέλουμε να συνεργαστούμε με τη Διεθνή Συμμαχία, με το Διεθνή Συναψηφισμό για να βρούμε τις ρίζες της τρομοκρατίας. Πιστεύουμε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή θα δημιουργήσει ακόμα πιο πολλές ακραίες ομάδες στη Συρία, την Ιεμένη ε, και αλλού, τη Λιβύη και αναζητούμε τις ρίζες της τρομοκρατίας για να εξασφαλίσουμε ασφάλεια Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μετριοπαθώς τη συνεργασία μας στην περιοχή, στη, την περιφερειακή συνεργασία δηλαδή. Θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας και τις άλλες περιοχές στην περιοχή μας. Είναι δύσκολη η, πρόκληση αυτή. Θα θέλαμε στο μέλλον να η συνεργασία να έχει θετική Ειδικά στοιχεία συνεισφοράς. Ε, θα θέλαμε να είμαστε μεταξύ των χωρών που θα ε, α, διευκολύνουν στην επίλυση των προβλημάτων. Ε, έχουμε κάνει βήματα πρόοδου με τη Σαουδική Αραβία, με την Τουρκία και με άλλους γειτονές μας. Θέλουμε οι διμερείς διαφορές να λύνονται ειρηνικά, αλλά πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα στην περιοχή μας, όχι μόνο για το Ιράκ, αλλά για όλη την περιοχή και την Ευρώπη. Και συνεργαζόμαστε με χώρες. Η συνεργασία αυτή θα μας βοηθήσει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ, η, συμφωνία αυτή θα, η συνεργασία αυτή θα μας βοηθήσει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια καινούρια συνεργασία σε θέματα περιβάλλοντος, υδάτινων πόρων, ε, οικονομίας και Επενδύσεων και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας. Χρειαζόμαστε βοήθεια για την ανοικοδόμηση, όχι μόνο για τις περιοχές που έχουν πιο πολύ πληγή, αλλά για όλη τη χώρα. Από το, 19, από το δεκαετία του 80 δεν έχει γίνει κάποια ανοικοδόμηση. Αυτό πρέπει να γίνει στο μέλλον λοιπόν. Ως κυβέρνηση του Ιράκ έχουμε ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα καινούριο περιβάλλον για να προσελκύσουμε ξένες εταιρείες και επενδύσεις. Δεν θα είναι εύκολο γιατί έχουμε διαρθρωτικά προβλήματα. Θα χρειαστεί χρόνος. Όμως η κυβέρνηση μπορεί ήδη να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις και να τις αρχίσει να τις υλοποιεί. το Ιράκ θα μπορούσε να γίνει σημείο εστίασης ε, για την δραστηριοποίηση στις χώρες της περιοχής και θα ήταν χρήσιμο να έρθουν οι Ευρωπαίοι να δουν την κατάσταση στο Ιράκ που είναι πολύ καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή Οι εκλογές που θα λάβουν χώρα σε δύο εβδομάδες θα δείξουν ε, ότι απομακρυνόμαστε από την σεκταριστική και εθνοτική βία. Προσπαθούμε να ξεφύγουμε από το διχασμό και ίσως αυτό αυτές οι εκλογές αποτελέσουν ε, μια καινούργια αφετηρία για την εσωτερική μας πολιτική. Ε, ίσως ο διχασμός δεν θα εξαλειφθεί αμέσως, αλλά οι επόμενες εκλογές θα αποτελέσουν ένα δείγμα γραφής για το μέλλον. Ε, οι εξελίξεις του Ιράκ είναι μοναδικές στον αραβικό κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα εκλογική και δημοκρατική. στη Βαγδάτη και στο Ιράκ ε, γενικά ο κόσμος έχει πολλές προσδοκίες για τους υποψήφιους. Ε, είναι πολύ σημαντικό να εγκαθιδρύσουμε το κράτος δικαίου ε, το οποίο έχει πληγεί από το 2003 από, την, ε, από τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ε, εκπαίδευση, καλύτερη εκπαίδευση των, ε, του στρατιωτικού μας προσωπικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη μας βοηθάει στην ε, ανάπτυξη ικανοτήτων τα τελευταία χρόνια. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι της συνεργασίας. Ελπι, ε, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποτελέσει και παράδειγμα ε, για τον, την πολιτική μας μετάβαση με τις αρχές της και τους κανόνες της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα στηρίζει την ακαιρεότητα και την ενότητα στο Ιράκ Και μαζί με την ανοικοδόμηση είναι πολύ σημαντικό ε, να εκπροσωπούνται και τα τοπικά συμφέροντα, οι τοπικές μειονότητες, ε, η Ραμάντη, η Σελαχαντίν, ε, οι θρησκευτικές μειονότητες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε αυτή την ενότητα. Η επόμενες εκλογές, οι επικείμενες εκλογές, θα είναι μια ευκαιρία. Ε, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούσαν το Σύνταγμά μας και την ενότητα του κράτους συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό επίσης οι εκτοπισμένοι να επιστρέψουν στις εστίες τους. Και αυτό συμβαίνει και είναι επίτευγμα και για την κυβέρνηση αλλά και για όλους όσους στήριξαν την επιστροφή, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Είναι μεγάλη η πρόκληση, αλλά είναι σαφές το προς τα που κινούμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Υπουργέ για τα πολύ σύντομα αλλά πολύ σαφή σχόλια σας. Έχουμε χρόνο για τη συζήτησή μας τώρα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Συνέχεια θα σας δώσουμε το λόγο για να απαντήσετε. Πρώτος ομιλητής ο Αρόντα Αρζάν για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την εισήγηση. Το Ιράκ εισέρχεται σε μια φάση σταθεροποίηση που είναι κρίσιμη και ελπίζουμε να είναι λιγότερο χαόδες από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Είμαι πεπισμένο λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει και χαιρετίζω ακριβώς την παρουσία σας εδώ για να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό η συνέλευσή μα να πάει επιτέλου στο Ιράκ. Είχαν γίνει προσπάθειες παλαιότερα, αλλά εμεί ήμασταν έτσι πιο διστακτικοί. Λυπάμαι βέβαια γι' αυτό και ελπίζω να έχουμε ευκαιρία να πάμε και ιδιαίτερα ελπίζω να είμαστε σε θέση να εργαστούμε σε θέματα διακυβέρνηση και ασφάλεια. Γιατί όπω είπατε και εσεί στο τέλο τη εισήγηση, τα εδάφη που έχουν ανακτηθεί από το Ισλαμικό κράτος και η διακυβέρνησή τους είναι σημείο κλειδί για την ε, παγίωση της σταθερότητα και την εξάλληψη των τρομοκρατικών ομάδων. Μια ερώτηση έχω παρ' αυτά για την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας που αναφέρατε ως ένα τομέα πιθανής συνεργασίας με ποια είναι η θέση μας. Δηλαδή, μήπως η θέση μας ήδη έχει καλυφθεί από τις ΗΠΑ και το Ιράν, έτσι, για να αναφέρω δύο σημαντικές χώρες που είναι έντονα παρούσες στο Ιράκ. Θεωρείτε λοιπόν ότι εμείς έχουμε θέση τη στιγμή που αυτές οι δύο μεγάλες χώρες ήδη καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο στα θέματα ασφάλειας και αν η απάντησή σας είναι καταβατική, τότε ποιος συγκεκριμένα θα ήταν ο ρόλος της Ένωσης που θα μπορούσε να διαδραματίσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντανζόν. Υπουργέ θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, διότι ένα από τα θέματα που μας ανησυχούν ιδιαίτερα είναι πώς μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανοικοδόμηση στις απελευθερωμένες περιοχές, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης και παροχής ευκαιριών απασχόλησης στους πολίτες μας μέσω της προσέλκυσης εταιριών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις. Και όταν μιλούμε για επενδύσεις θεωρούμε ότι είναι μια πραγματική ευκαιρία για την ανοικοδόμηση του ε, Ιράκ, διότι στην διαδικασία σταθεροποίησης της χώρας ε, ένα από τα βασικότερα ζητούμενα είναι η ανοικοδόμηση και η παρουσία ξένων εταιρεών ε, για την οικοδόμηση αυτοκινητοδρόμων, σχολείων, νοσοκομείων είναι μια διάσταση εξαιρετικά σημαντική. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κρίσιμος. Γιατί δεν υπάρχουν μεμονωμένε χώρε που μπορούν να προσφέρουν αυτό που μπορεί να μα προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν η ΕΠΑ. Όταν μιλούμε για τη δημιουργία ικανοτήτων, ε, ε, όταν μιλούμε για ανθρώπινα δικαιώματα και την εφαρμογή και την υποβολή του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση από την κυβέρνηση. Αυτά τα στοιχεία, αυτές οι διαστάσεις είναι πολύ σημαντικές. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποστήριξη της μετάβασης προς τη δημοκρατία διαφόρων χωρών είναι πολύ σημαντικός. Και νομίζω ότι καμία μεμονωμένη χώρα δεν μπορεί να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο μόνη της. Ε, πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδωσε και κίνητρα για να προβούμε σε μεταρρύθμιση στον τομέα της ασφάλειας ε, και, την μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεών μας. Ε, και αυτή τη στιγμή μια τέτοια διαδικασία βρίσκεται υπό εξέλιξη. Βρίσκεται σε διαδικασία ε, σε, σε εξέλιξη μια φάση οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Θεωρώ επίσης ότι η εκπαίδευση δικαστών και η παροχή ευκαιριών προς αυτούς, ε, προκειμένου να εφαρμόζουν το κράτος δικαίου, είναι κρίσιμη σημασία για το Ιράκ. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή, αξιοποιώντας και την ειδική σχέση που έχει με γειτονικέ χώρες. Και εμείς ήδη έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτό που πιστεύουμε πραγματικά είναι ότι η έννοια της συνεργασίας είναι, είναι καινούρια στην περιοχή. Υπήρχε πάντοτε ένας ανταγωνισμός ε, μεταξύ των χωρών της περιοχής. Ε, κάθε χώρα προσπαθούσε να επιβάλλει το δίκαιό της ε, και μάλιστα με λάθος εργαλεία. Δεν επέλεγαν στο παρελθόν οι χώρες της Μέσης Ανατολής τη συνεργασία την, στον οικονομικό τομέα στις επενδύσεις για παράδειγμα. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ καινούρια για εμάς. Γι' αυτό χθες ε, αποστήλαμε και επίσημη πρόσκληση προς τις ε, γειτονικές μας χώρες προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα, ε, στην ηλεκτρική ενέργεια. Εμείς στο Ιράκ φυσικά θέλουμε στο Ιράκ επίσης να υπερβούμε και τον θρησκευτικό διχασμό. Ε, δεν θέλουμε να μπούμε στη μέση ε, ανάμεσα στον, στον ανταγωνισμό που υπάρχει μεταξύ Κατάρ και Τουρκίας για παράδειγμα. Θεωρούμε ότι η κρίση που μαστίζει την περιοχή μας πρέπει να επιληθεί με ειρηνικά μέσα. Δεν θέλουμε κλιμάκωση ούτε στη Συρία ούτε στην Ιεμένη. Δεν θα φέρει τίποτα κάτι τέτοιο. Βλέπουμε τη βία τα τελευταία έξι χρόνια. Και το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι χωρίς πολιτική συμφωνία δεν μπορείς να επιτύχεις τίποτα. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να εμπλακεί στην ε, διαδικασία και στην κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή. Γιατί βλέπουμε ριζοσπαστικοποιημένους, ε, τρομοκράτες, πρόσφυγες, όλα αυτά είναι θέματα που αφορούν άμεσα και την ε, Ευρώπη λόγω και της γεωγραφικής μας εγκύτητας. Ίσως όχι τόσο της, της για παράδειγμα. Για, για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει το Ιράκ, την Τινησία και άλλες χώρες που με σοβαρότητα καταβάλουν προσπάθειες για μια μεταρρύθμιση και μετάβαση. Υπάρχουν λοιπόν ήδη ε, πολλά παραδείγματα υποστήριξη που έχουμε λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε, είμαστε πολύ ευγνώμονες και θέλουμε αυτέ οι προσπάθειε και από τι δύο πλευρέ να συνεχιστούν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Συνάδελφοι, υπάρχει κάποιο άλλο που θα ήθελε να θέσει ερωτήματα ή να κάνει κάποια παρατήρηση, παρέμβαση στη συζήτηση. Όχι από ό,τι βλέπω. Κύριε Υπουργέ, θέλετε να μας πείτε κάτι ακόμη. Θα ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε σήμερα και να εκφράσω την ελπίδα μου ότι θα υπάρξει και μια επίσκεψη της Επιτροπής σας στη χώρα μου. Είστε ευπρόσδεκτοι οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Πρόεδρος, κύριε Υπουργέ, σας υπόσχομαι ότι ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχουμε πρόθεση να πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στο Ιράκ. Σκεφτόμαστε, σχεδιάζουμε να κάνουμε μια τέτοια επίσκεψη ε, κατά πάσα πιθανότητα το Δεκέμβριο. Φυσικά χρειάζεται να περάσουμε και από, από ελέγχους ασφαλείας κτλ. Αυτός όμως είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η πρόθεσή μας και ε, προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με όλους τους ε, συνομιλητές και να εκφράσω και εγώ από αυτό το βήμα την απόλυτη προσήλωσή μας προς το στόχο της ανοικοδόμησης του Ιράκ. Ας ελπίσουμε λοιπόν να γίνει αυτό το ταξίδι, αυτή η επίσκεψη το Δεκέμβριο. Άρα, αφού δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία του εδώ ε, και θα αναστείλουμε την ε, συνεδρίασή μας. Θα συνεχίσουμε στις 2.30 με το εργαστήριο με θέμα της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Ευχαριστώ.